Um, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Σε αυτήν την τόσο σημαντική ακρόαση που έχουμε όσον αφορά τις συμφωνίες για συνεργασία με τρίτες χώρες σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης και τις επιστροφές. Έχουμε εδώ και την Επιτροπή Ανάπτυξης, της οποίας ε, τα μέλη είναι εδώ, ο πρόεδρος είναι σε αποστολή και λείπουν και κάποια μέλη από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Είμαστε εδώ κυρίως μέλη της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ. Να ξέρετε ότι αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο συνεδρίαση αυτή και μπορείτε να την βρείτε στην ε, ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος της σημαντικής αυτής ακρόασής μας σήμερα είναι να εξετάσουμε στοιχεία κλειδί της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες όσον αφορά τη διαχείριση τη μετανάστευση. Και αυτό προκειμένου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούσει τις απόψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των Ακαδημαϊκών και των διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ. Να ξέρετε ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τα Δανέζικα, τα Μαλτέζικα, τα Κροατικά και τα Γκέλικ. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή εισαγωγή για να έχουμε χρόνο να ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας. Λοιπόν, θα χωριστεί σε τρία τμήματα, σε τρία πάνελ η σημερινή συζήτηση. Το πρώτο θα ασχοληθεί με τη συνεργασία μας με τρίτες χώρες τις δημοκρατικές αρχές, πώς ε, τηρούνται κλπ. Το δεύτερο πάνελ θα ασχοληθεί με τις εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας ε, που έχουμε και αποτελούν μέσω διαλόγου και συνεργασίας με τρίτες χώρες. Το τρίτο πάνελ θα ασχοληθεί με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιστροφές. Η εξωτερική διάσταση Τη ε, πολιτική μετανάστευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικεντρώνεται στη συνεργασία με τρίτε χώρε για να αντιμετωπιστούν οι ρίζε τη μετανάστευση και να αντιμετωπιστούν επίση και οι παράτυπε ροέ προ την Ευρώπη. Η συνεργασία, οι εταιρικέ σχέσει με τι χώρε προέλευση, transit και ε, προορισμού αποτελούν στοιχείο κλειδί για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πάνελ ευθύς που έχει να κάνει με την μετανάστευση ε, πλαίσιο εταιρική σχέση και ενίσχυση τη συνεργασία. Πρώτο μα ο είναι ο Λεωνέλο Καμπρίτσι που είναι τμήματάρχη για την ε, μετανάστευση και την ε, ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής δράση. Έχετε το λόγο παρακαλώ για 10 λεπτά κύριε Καμπρίτσι. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. 10 λεπτά. Ωραία. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ παρόλο που έχω πολλά να σας πω και κατά πάσα πιθανότητα θα σας πω πολλά πράγματα έτσι πολύ βιαστικά σαν καρικατούρα κάπως και ίσως δημιουργηθεί και σύγχυση γι' αυτό και θα αρχίσουμε τα συμπεράσματα πριν περάσω για να καταλάβετε γιατί σας λέω αυτό που σας λέω. Και ποιο είναι το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί η μετανάστευση, η μετακίνηση των ανθρώπων, πληθυσμών είτε είναι πρόσφυγες είτε όχι, χωρίς να έχουμε μια αξιόπιστη εξωτερική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να χτίσουμε για τη μετανάστευση από μόνοι μας. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες, είτε είναι χώρες προέλευσης είτε transit και θα σας πάρουν στα σοβαρά μόνο αν είσαστε σοβαροί σε αυτά που έχετε να τους προσφέρετε. Αν απλώς τους στέλνετε πίσω και τους λέτε να λύσει συνεργασία από εδώ, λίγο από αυτό, λίγο από εκείνο, δεν θα καταλήξετε πουθενά. Αυτό το οποίο χρειάζεστε, είσαστε εταίρους που να αντιλαμβάνονται ότι ανεξάρτητα από το θέμα της Ευρώπης, της μετανάστευσης, έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστιες προκλήσεις και πρέπει να βρουν το δικό του μοντέλο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξη που είναι βιώσιμο μέσα σε, ένα, μέσα σε μια παγκοσμιοποίηση που έχουμε σήμερα. Και μόνο έτσι θα καταφέρετε να διαχειριστείτε την μετανάστευση. Λοιπόν, θα προσπαθήσω τώρα κάπως σύντομα να σας εξηγήσω γιατί το βλέπω έτσι, γιατί σας στέλνω αυτό το μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, κάπως σύντομα, θα δω χρονολογικά και ιστορικά τις δύο τάσεις που έχασε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να έχει αξιόπιστη μεταναστευτική πολιτική απέναντι σε τρίτες χώρες. Τώρα είμαστε στην τρίτη ευκαιρία μπροστά, ελπίζω να μην τη χάσουμε κι αυτή. Θα σας υπενθυμίσω ότι έγινε στις 11 Σεπτεμβρίου στις Ηνωμένε Πολιτείες και από τότε ξεκίνησε η σταυροφορία κατά της τρομοκρατίας σε όλη τη Μέση Ανατολή, Αφγανιστάν, Πακιστάν κτλ. Σας τα λέω βιαστικά όντως. Κάποια στιγμή οι ευρωπαϊκές χώρες είχαν, μπήκαν στον πειρασμό μάλλον να ακολουθήσουν αυτή την σταυροφορία με τις συνέπειες που γνωρίζουμε και με την πολιτική για τις χώρες γειτονίας που αναπτύξαμε το 2003-2004. Είχαμε αρχίσει και ενισχύθηκε αυτή αργότερα. Μετά είχαμε το φαινόμενο των σχεδιών που περνούσαν από την Αφρική στην Ισπανία. Η ευκαιρία που χάσαμε ήταν ότι δεν χρησιμοποίησαμε την πολιτική γυτνίαση με τη σωστή μερίσια διάταξη ώστε να δούμε την εξωτερική διάσταση της κοινοτική πολιτικής, να έχουμε συμφωνίες είτε για την έρευνα, είτε για τη γεωργία, είτε για οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί ο νους του ανθρώπου και να τα χρησιμοποιήσουμε σαν εξωτερική διάσταση των κοινοτικών μας πολιτικών μέσα σε ένα πακέτο ευρωπαϊκό για να ανταποκριθούμε στο αίτημα τρίτων χωρών και μέσα σε αυτό το θεματολόγιο να βάλουμε και κάτι για την κοινή από κοινού αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του μεταναστευτικού γενικότερα. Αποτύχαμε λοιπόν σε αυτή την ευκαιρία, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Και όχι γιατί ήταν κακή η πολιτική γειτονία, αλλά γιατί για να δουλέψει η πολιτική αυτή θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πιο σοβαρά τις χώρες που είχαμε απέναντί μας και να φροντίσουμε να έχουμε τη στήριξη όλων των χωρών μελών. Και τι διαπιστώσαμε ήταν ότι κάποιες χώρες, ή την Ιγυρία με αλλά όχι μόνο, εντάξει μπορεί να μην ήταν ο πιο κατάλληλος εταίρος, αλλά πάντως από τη δικιά μας την πλευρά, από την άλλη, εξακολουθούμε να έχουμε χώρες οι οποίες εξακολουθούν να βάζουν προτεραιότητες ε, λάθος στις σχέσεις μας με τις τρίτες χώρες. Βάζουν, προτάσουν δηλαδή το διμερές αντί να προτάσουν το συλλογικό, δηλαδή τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό δεν λειτουργήσε λοιπόν αυτή η ευκαιρία. Το δεύτερο τρένο που χάσαμε ήταν μετά την Αραβική Άνοιξη. Δεν έχουμε πια τον Πέναλι. Και τι κάναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πήγαμε να δούμε όλες αυτές τις χώρες με το σύνθημα More for More, περισσότερα για περισσότερα. Το ανόητο αυτό το βάζω εισαγωγικά, έτσι, περισσότερα για περισσότερα. Γιατί όσο περισσότερο δημοκρατικοί γίνεστε, θα έλεγα εγώ, όλο και περισσότερη συνεργασία θα σας δώσω. Δεν λειτουργεί και δεν λειτουργήσε. Οπότε είχαμε την ευκαιρία να το κάνουμε ανάποδα. Δηλαδή, όσο περισσότερα εσείς αποφασίζετε να συνδέσετε δηλαδή το δικό σας οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο με την Ευρώπη, την εσωτερική μας αγορά κτλ. Τόσο περισσότερα θα σας ζητήσω κι εγώ να ασπαστείτε τις δικές μας αξίες, κράτος δικαίου κτλ. Και τότε γινόμαστε εταίροι. Δεν δίνουμε απλώ μαθήματα. Και αυτό ήταν το δεύτερο τρένο που χάσαμε. Και έρχομαι στο τρίτο, και με αυτό θα τελειώσω. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι η μεταναστευτική κρίση, όπως ονομάστηκε, που ουσιαστικά ήταν ε, προσφυγική από τη Συρία κρίση, οι κρίσεις αυτές ήταν στα πρωτοσέλιδα όλων των εφημερίδων και ανάγκασαν τις χώρες μέλη να αντιδράσουν και αντέδρασαν με τη διάσκεψη των Βαλκανίων, της Βαλέτα, ένα σωρό ωραία πράγματα. Δουλέψαμε και εμείς με αυτά, είναι σημαντικά, όμως παρόλα αυτά το πρόβλημα παραμένει το ίδιο. Αν Τώρα έχουμε το πλαίσιο εταιρική σχέση που είναι η ιδέα το κατά πόσο έχουμε μια πραγματικά διμερή σχέση με πραγματικά κοινό θεματολόγιο κτλ. Ε, λοιπόν, τώρα αυτό πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο τρένο, η τρίτη ευκαιρία που ελπίζουμε να μην χάσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πραγματικά από κοινού έχουν ε, προτείνει ό,τι μέσα και εργαλεία ε, μπορούσαν να προτείνουν και έχουν μια αντιμετώπιση αναχώρα, γιατί για την κάθε χώρα χρειαζόσαστε αρρωγή, χρειάζεστε ειδική αντιμετώπιση, εταιρική σχέση και συνολική εικόνα 360 μοιρών. Πρέπει να είμαστε σε θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρουμε περισσότερα πράγματα συλλογικά από όσα θα μπορούσε κάθε χώρα χωριστά. Είτε πρόκειται για την κοινή γεωργική πολιτική, τη γεωργία δηλαδή, είτε πρόκειται για άλλα. Συνολική προσέγγιση. Και τέλος υπάρχει και το Ευρωπαϊκό ε, Σχέδιο Στρατηγικών Επενδύσεων που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για συνεργασίες και για επενδύσεις στις χώρες αυτές. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για χρήματα από τις αναπτυξιακές βοήθειες που θα δώσετε, που δεν φτάνουν έτσι καλλιώς, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Πρέπει να μπορούμε να επενδύσουμε σε χώρες που είναι διατεθειμένες να παίξουν το παιχνίδι, που είναι διατεθειμένες να ενηλικιοποιηθούν μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Μόνο έτσι θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, μεταξύ άλλων, και η πρόκληση της ηρεμίας, προκειμένου ο δικός τους ο πληθυσμός να αποκτήσει αυτά που χρειάζεται. Θα σταματήσω εδώ, νομίζω ότι μακρηγόρησα έτσι καλλιώς. Και από εκεί και πέρα αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστως τότε να συζητήσουμε περισσότερο την τρέχουσα κατάσταση και εν ώψη μάλιστα τη διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική, αλλά και τη σχέση μα με τη Λιβύη, που αποτελεί μια προτεραιότητα για μα. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ συνθετικά μα τα είπε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Εντάξει, τα είπατε συνοπτικά, αλλά πολύ ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενος, επόμενη ομιλήτρια για θέματα που αφορούν περισσότερο την Αναπτυξιακή Επιτροπή για την ε, ε, πολιτική και θα μας μιλήσει εκ μέρους της Κάριτας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Μποντό. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω την άποψη της κοινωνίας των πολιτών για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα λοιπόν θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη, μια καλύτερη προσέγγιση σχετικά με τη δυνατότητα μετακίνησης των ανθρώπων. Εμείς η Κάριτας είμαστε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, έχουμε 49 οργανώσεις μέλη, ε, Είμαστε παρόντες σε 160 χώρες, προσφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια και συνεργασία για θέματα ανάπτυξης. Ε, πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμεθα δημιουργήθηκε λόγω της ε, κρίσης ε, του προσφυγικού. Ε, καλύτερα όμως να μιλήσουμε για κρίση αλληλεγγύης και εσωτερικής πολιτικής κρίση αλληλεγγύης προς τρίτες χώρες. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το 85% των προσφύγων ανά τον κόσμο φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και αν δείτε μια χώρα όπως η Ιορδανία, κάθε έκτος πολίτη στην Ιορδανία είναι πρόσφυγας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι οι τρίτες χώρες κάνουν πάρα πολλά για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ε, μετανάστευση οδήγησε στο να αναζητήσουν πολιτική τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ε, θέλησαν να συζητήσουν με τρίτες χώρες ε, για να διαχειριστούν το προσφυγικό και ενδεχομένως και να αναχαιτήσουν τις ε, μεταναστευτικές ροές. Αυτό το πλαίσιο συνεργασίας σημαίνει συνεργασία με τρίτες χώρες με στόχο να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα στόχοι που αφορούν στο μεταναστευτικό. Βλέπουμε όμως ο βασικότερος στόχος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αυξηθούν οι επιστροφέ και οι συμφωνίες επαναπρόθεσης. Πέντε αφρικανικές χώρες αδιαφορούν Νιγηρία, Νίγηρα, Μαλή, Σενεγάλη και Αιθιοπία. Αυτές είναι πέντε χώρες με τις οποίες ε, έχουμε συζητήσει και διαπραγματεύσει. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο συνεργασίας έθεσε αρκετές ε, προκλήσεις ε, αλλά και ερωτηματικά το πρώτο είναι ε, το θέμα της ασφάλειας. Η εσωτερική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη μετανάστευση κυριαρχεί σε αυτή την εταιρική σχέση. Ε, στόχος είναι ελεγχή στα σύνορα, να αναχαιτιστούν οι μεταναστευτικές δουλειές και να υπάρξουν περισσότερες επιστροφές σε τρίτες χώρες. Αυτό είναι ένας βραχυπρόθεσμος στόχος που έχει σχέση με το να μπορούν να πούν οι πολιτικοί στα μέσα ενημέρωση ότι έχουν αναχαιτήσει τις ροε. Αλλά όταν προσπαθεί κανείς να αναχαιτήσει κάποιες ροέ, ε, θα ανοίξουν άλλε, θα προκύψουν άλλες και αυτό θα ενθαρρύνει άλλους διακινητέ ε, και άλλα δίκτυα. Ε, Επίση, να πούμε ότι οι αφρικανικές χώρες αυτές ενδιαφέρονται για αυτή τη συνεργασία και με χαρά άκουσα προηγουμένως ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταθέσει κάτι που να είναι σημαντικό για τις αφρικανικές χώρες, να θέλουν και εκείνες να συνεργαστούν. Γιατί αυτή τη στιγμή τα συμφέροντά τους δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι περισσότερες εξ αυτών δεν ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν τη μετανάστευση, το μεταναστευτικό. Σε Νεγάλη, πάνω από 13% του ΑΕΠ ε, προέρχεται από εμβάσματα τα οποία στέλνουν με οι μετανάστες τους στο εξωτερικό με βάση τα στοιχεία της ΟΝΤΙΡ. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να εξευρεθούν ε, ασφαλείς ε, τρόποι και δυνατότητες να μπορούν οι μετανάστες να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρομαι σε διευκολύνσεις για τη θεώρηση ή για άδειε εργασία. Πολλοί εμπειρογνώμονε έχουν θέσει το ερώτημα σε ποιο βαθμό αυτές οι συνεργασίες είναι πραγματικές συνεργασίες ανάμεσα σε δύο εταίρου που είναι και ισότιμοι. Επόμενη διαφάνεια. Η συνεργασία για θέματα ανάπτυξης ε, χρησιμοποιείται στην εταιρική αυτή σχέση ως ε, μια δυνατότητα μόχλευσης για να συνεργαστούν ε, οι τρίτες χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τις δικές της όμως προτεραιότητες. Άρα δηλαδή υπάρχουν θετικά και αρνητικά κίνητρα τα οποία χρησιμοποιούνται για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ότι θα υπάρχουν συνέπειες για όσους δεν θέλουν να συνεργαστούν ξεκινάμε από την παραδοχή ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα αναχαιτήσει τη μετανάστευση, οι οικονομικές δυνατότητες θα αναχαιτήσουν τη μετανάστευση. Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει ότι συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι έχουν περισσότερα οικονομικά μέσα, θέλουν περισσότερο να μεταναστεύσουν και ε, έτσι να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα το να χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια ως, ε, δυνατός, ως δυνατότητα μόχλευσης, ε, ίσως αυτό να αφορά περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ε, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ένα άλλο στοιχείο που δημιουργεί προβλήματα κατά την άποψή μας είναι ότι και τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα σε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις γιατί γίνονται διαπραγματεύσει με χώρες οι οποίες ε, δεν έχουν καλό ιστορικό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και επίσης λείπουν και οι σταθεροί μηχανισμοί σε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις. Παράδειγμα η συνεργασία με τη Λιβύη που πιο προκληματική σχέση. Η περίπτωση του Νίγηρα ε, πολύ συχνά ε, χρησιμοποιείται για να ε, αποδειχθεί ότι είναι επιτυχημένη συνεργασία, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Οι εμπειρογνώμονες στην περιοχή αμφισβητούν το γεγονός ότι στον Νίγηρα η στόχευση σε διαχείριση, στη διαχείριση του μεταναστευτικού ε, δεν προσφέρει όμως ε, πραγματικές οικονομικές δυνατότητες ε, στους νέους γιατί αυτοί πέφτουν στα χέρια εγκληματικών συμμοριών. Επίσης, ο έλεγχος στα σύνορα αυτός οδηγεί στο να αναζητούν οι ενδιαφερόμενοι νέες οδούς ε, πολύ επικίνδυνε. Για να ολοκληρώσω, ένα από τα προβλήματα σε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις είναι το γεγονός ότι αυτή η προσέγγιση εστιάζει κυρίω στην ασφάλεια και στις ε, επιστροφές. Ε, με τον τρόπο όμως αυτό υποσκάπτεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το επιβεβαιώνει και η έκθεση μιας επιτροπής της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ ότι η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνεται βράχει πρόθεσμα, μπορούμε όμως να εστιάσουμε μόνο σε θέματα ασφάλειας, να προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε τη μετανάστευση αντί να της δώσουμε νέα μορφή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι και οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες, σε μακροχρόνια προοπτική. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ισορροπημένη σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να είναι έτοιμη ε, να προσφέρει και κάτι το θετικό για τις χώρες τις οποίες συνεργάζεται, δηλαδή ασφαλή και νόμιμη μετανάστευση που θεωρητικά θα πρέπει να υπάρχει στο πλαίσιο συνεργασίας, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει. Ολοκληρώνω ε, με μια συγκεκριμένη σύσταση που αναφέρεται στην ε, προαγωγή του στόχου 17 που αναφέρεται στη διευκόλυνση της ε, μετανάστευσης, στη διευκόλυνση ε, των ε, μεταναστευτικών θεωρήσεων και των θεωρήσεων για σπουδές. Άρθρο 108 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Εκεί αναφέρεται ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για να αντιμετωπιστεί η φτώχεια. Επίσης αναφέρεται ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, σε σχέση με τις ε, τρίτες χώρες, να υπάρχει αυστηρός ε, μηχανισμός ελέγχου και να διασφαλίζεται επίσης ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες δεν σημαίνει την μείωση της ευθύνης ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα δικαιώματα των μεταναστών. Νομίζω επίσης ότι όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι βουλευτές πρέπει να συμμετέχουν σε διαδικασίες ελέγχου. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτές τις συμφωνίες ε, συνεργασίες. Και τέλος πιστεύω ότι ως πολιτικοί έχετε και την υποχρέωση να ευαισθητοποιήσετε τους πολίτες το τι ακριβώς σημαίνει μετανάστευση. Γιατί οι περισσότερες πολιτικές σημαίνουν αρνητικά στοιχεία, αναφέρουν ότι πρέπει να αναχαιτιστούν οι μεταναστευτικές ωραίες. Αυτό οφείλεται όμως στο ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι είναι μετανάστευση, δεν γνωρίζουν γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν. Άρα είναι θετικό να προβάλλονται θετικότερα στοιχεία όσον αφορά στη μετανάστευση. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταία <clears throat> ομιλήτρια που θα λάβει το λόγο στο παρόν πάνελ είναι η κυρία Μορένο Λάξ, η οποία είναι καθηγήτρια στο ε, Πανεπιστήμιο του Queen Mary στο Λονδίνο, στην νομική σχολή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με την άδειά σας θα παρουσιάσω την ανάλυση μου για το δίκτυο συνεργασίας για τη μετανάστευση και το έργο και το αποτέλεσμα του δικτύου αυτού. Το MPF, όπως είπε ένας αξιωματούχος ε, της Κομισιόν, είναι το καινούριο καλούπι για τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως είπε ο συνάδελφος ε, της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων, ε, μέσα στα πλαίσια του More for More και συζητεί το γράμμα, το πνεύμα, την πρακτική και τον απολογισμό του MPF έως τώρα. Παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια. Σύμφωνα με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που πρότεινε τη δημιουργία του MPF, στοχεύει στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μέσω σε βάθος συνεργασιών με τις ε, τρίτες χώρες. Και μιλούν για τον εκδημοκρατισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη των χωρών προέλευσης και διέλευσης με αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων στις ρίζες τους. Ταυτόχρονα μια συνολική προσέγγιση για την κινητικότητα και τη μετανάστευση, βραχυπρόθεσμες δράσεις, αντιμετώπιση της λαθροδιακίνησης, και ενίσχυση των επανεισδοχών. Αυτά λέει το γράμμα του MPF. Για το πνεύμα τώρα του MPF και αντίθετα με την συνολική προσέγγιση για τη μετανάστευση και κινητικότητα και σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουνίου του 2016 στοχεύουν στην πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και σας λέω όπως τα λέει το κείμενο της συμπερασμάτων του Συμβουλίου, που θα γίνει με οποιοδήποτε μέσον στην πράξη, με ε, προσωρινές ανεπίσημες ε, ρυθμίσεις, με χρήση κάθε αποτελεσματικού κινήτρου ή επιβολής όρων, είτε με αναπτυξιακή βοήθεια είτε μέσω του εμπορίου, ανεξαρτήτως των αρχικών στόχων τη ε, πολιτική αυτής όπως είπε και η συναδελφό μου της ε, Κάριτας και αναζητώντας συνέργειε με τις χώρες μέλη με διμερείς ενέργειες με άλλους εταίρου, Τουρκία, Λιβύη, όποιε και αν είναι οι επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτικών των χωρών αυτών. Έρχομαι τώρα στην πρακτική. Τι σήμανε το MPF επιτόπου. Μέσα στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της κεντρικής οδού της Μεσογείου Ήδη από το καλοκαίρι του 2015 το MPF έχει υλοποιήσει του στόχους του μέσα από μια σειρά δράσεων που μεταφέρουν το πνεύμα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου που ανέφερα προηγουμένω στο ε, πεδίο. Με προγράμματα όπως UNAFORMED, το τρίτο EUBAM που είναι η αποστολή στη Λιβύη και που έχουν κινητοποιηθεί για να ενισχύσουν την ικανότητα των ε, Λίβιων να ανακόψουν τα ανεπιθύμητα ρεύματα. Έχουν δαπανίσει άνω των 100 εκατομμυρίων ε, ευρώ, μεταξύ άλλων από το Ταμείο για την Αφρική, για να βελτιωθούν τα κέντρα συγκέντρωσης και υποδοχής στην Λιβύη, να ενισχύσουν τις, ε, την, εκπαίδευση των λιβικών δυνάμεων και το καθεξής. Οι δε Ιταλοί έχουν συμβάλει και πολιτικά και οικονομικά στην προσπάθεια αυτή μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νέος κώδικας ε, δεοντολογίας που εγκριθήκε, καθώς και το Μνημόνιο Συμφωνίας για την κυβέρνηση της Βενγκάζης αλλά και με τις πολιτοφυλακές και σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση των ΗΠΑ του Ιουνίου 2016 ενισχύουν την ε, δράση της Ένωσης για την επίτευξη των στόχων του MPF. Για τους μετανάστες αυτή η συντονισμένη παρέμβαση σημαίνει ότι έχουν ε, αποκλειστεί σε θύλακους, σε θύλακους μάλλον, απίστευτης με, ε, όπου δεινοπαθούν απίστευτα. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορώ να σας τα παρουσιάσω αυτά, αλλά θα ήθελα να τα παρακολουθήσετε με, τη, με την ησυχία σας στην, στο σύνδεσμο που σας δείχνω. Συνεργασία μεταξύ Ιταλικού Ναυτικού, ε, Λιβικής Ακτοφυλακής και του κέντρου της Ρώμης σε μια ε, επιχείρηση pullback που παρουσιάζονται ως δίθεν επιχειρήσεις διάσωσης και που αναλαμβάνονται από τη Λιβύη μετά από αίτημα ή εντολές της Ιταλίας και επειδή η Λιβύη δεν έχει δική της ζώνη έρευνας και διάσωσης, δεν έχει κέντρο συντονισμού των προσπαθειών διάσωσης δικό της, ούτε έχει και τις σχετικές ικανότητες δικές της η Λιβύη με κανένα τρόπο επίσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές μέρος για ευάλωτα άτομα που σύμφωνα δηλαδή με τις ε, ναυτικές συμβάσεις Maritime και Σόλας. Αυτά γίνονται με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πάντως χωρίς ε, ευθεία καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών μελών της. Αυτέ οι άμεσε διασυνδέσεις δηλαδή μεταξύ Ιταλικών αρχών και τη Λιβικής ακτοφυλακή και η φύση των κοινών παρεμβάσεων δείχνουν την άμεση συμμετοχή της Ιταλίας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δράσεις οι οποίες θέτουν τους ε, μετανάστες σε σοβαρό κίνδυνο σοβαρών παραβιάσεων των ε, ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Σύμφωνα με τα άρθρα για την ευθύνη των κρατών της Διεθνούς Σύμβασης και που έχουν σχέση και με το εθνικό δίκαιο και του κώδικα ανθρώπινων δικαιωμάτων, ερμηνείας ανθρώπινων δικαιωμάτων του Στρασβούργου και τις σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου. Ο απολογισμός των εργασιών του MPF λοιπόν είναι στην πραγματικότητα εξαιρετικά φρικτός. Έχει αλλάξει την ε, φύση της πολιτικής, οδηγεί σε αποδημοκρατισμό για την συγκράτηση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Δεύτερο, οι εξωτερικές σχέσεις έχουν λάβει πλέον άτυπη μορφή μέσω ε, συμφωνιών, μέσω μνημονίων, συνεργασία, μνημονίων συνεργασίας και ούτω καθεξής που βρίσκονται μέσα στο κέντρο, στον πυρήνα του MPF με αυτά τα συνολικά πακέτα τα οποία, στα οποία συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λιβύη αλλά και με άλλες χώρες τα οποία ξεφεύγουν από τον δημοκρατικό έλεγχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει φωνή, Εννοείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει φωνή, δεν έχει τίποτε να πει. Το άρθρο 16 της, ε, της ε, συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παραγκονιστεί. Τρίτο, δεν υπάρχει τρόπος πραγματικής παρακολούθησης ελέγχου για το πώς διατίθενται οι πόροι, τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτών. Δεν γνωρίζουμε εάν τα χρήματα αυτά πηγαίνουν για χρηματοδότηση δράσεων παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή για αντιμετώπιση των ε, δικτύων λαθροδιακινητών που υποτίθεται ότι καταπολεμεί το MPF. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, νομικές δεσμεύσεις, αυτές υποσκάπτουν τις ε, αρχές του διεθνούς δικαίου. Στην πραγματικότητα, δεν περιλαμβάνονται στις συμφωνίες αυτές. Και αυτό αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατιμορρησίας. Για αυτό η σύστασή μου είναι να επιστρέψετε στο αβ των εξωτερικών σχέσεων και στις αρχές που έχουν εμπνεύσει την ίδρυση την ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε το άρθρο 21 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή θα είναι μια πολύ καλύτερη επένδυση στην πραγματικότητα, θα οδηγήσει στην επιστροφή στη δημοκρατία, στο κράτος δικαίου, στην τόνωση των, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην αλληλεγγύη και, στην, και στο σεβασμό των ίδιων των αρχών του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνεται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Αν σας ενδιαφέρει η πλήρης ανάλυση σας παρακαλώ να εξετάσετε τους δύο συνδέσμους που βλέπετε στην διαφάνεια και αντίγραφα των δύο κειμένων είναι διαθέσιμα για τα μέλη της Επιτροπής σας μέσω της Γραμματείας της Επιτροπής Θεμεριδών Ελευθεριών. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε αμέσως τώρα στα μέλη. Δύο-τρία λεπτά παρακαλώ η κάθε παρέμβαση. Βέβαια, σας αντιλαμβάνομαι ότι όλοι θέλετε να μιλήσετε. Δύο-τρία λεπτά όπως είπα. Η κυρία Σοφίντ Φέλτ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη γιατί τα περισσότερα που ήθελα να πω τα είπανε η κυρία Μορδέ και η κυρία Μορένου Λάξ. Νομίζω ότι τέλεια εκθέσατε την κατάσταση με μία μικρή προσθήκη. Ξεχνάμε όταν ο κόσμος λέει ότι είναι εύκολο να κάνει κάνει συμφωνία με τη Λιβύη, να στείλει χρήματα στη Λιβύη, Μα έγινε και πριν από δέκα χρόνια από τον Περλουσκόνη. Και με τη στήριξη της ευρωπαϊκή Ένωσης έγινε συμφωνία με τη Λιβύη, ούτε και αυτό λειτουργήσε. Οπότε το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στους αυτούς μας πρόεδρε είναι πώς θα κάνουμε έναν ελάχιστο έλεγχο. Χτες το απόγευμα θύμωσα έχουμε τέτοιες συναντήσεις ξανά και ξανά και ξανά έρχεται ο ένας έρχεται ο άλλος και εξορχιζόμαστε. Μα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε πλήρως τις δυνάμεις μας, τα μέσα που έχουμε στην διάθεσή μας για να κάνουμε κάποια κάποιο ουσιαστικό έλεγχο στα θέματα του προπολογισμού που είμαστε εμείς ε, αρμόδιοι. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι μέλη σέβονται τις συνθήκες και κάνουν όντως πρόοδο όσον αφορά το κοινό σύστημα ασύλου, αντί να βρίσκουμε έτσι διάφορες παρακαμπτικές ε, οδούς. Γιατί τελικά αυτό κάνουν, αυτό γίνεται και λυπάμαι που το λέω. Υπάρχουν όλες αυτές οι συμφωνίες, οι οποίες είναι εκτός συνθήκων. Ενώ έχουμε νομικά μέσα στη διάθεσή μας οι χώρε μέλη αρνούνται να τα χρησιμοποιήσουν και ανταυτού βρίσκουν ε, διάφορες δεξιόδους δεξιά και αριστερά. Τι θα κάνουμε λοιπόν πρόεδρε, θέλω να ακούσω, να μάθω τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας και πώ θα τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα πράγματα γίνονται και ρυθμίζονται όπως πρέπει, ότι θα επιστρέψουν μέσα στα πλαίσια των συνθηκών και δεν θα παραμένουν εκτός. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη τώρα. Ευχαριστώ πολύ τους ε, συγητές ε, και κυρίως ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βιολέτα Μορένο Λάξ και την εκπρόσωπο της Κάριτας που μας έδωσαν πάρα πολλές και χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Τι σημαίνει επιτυχημένη εξωτερική πολιτική με βάση αυτά που είπε ο κύριος Γκαμπρίτσι. Εγώ έχω την εξής άποψη ότι αυτές οι πολιτικές επιστροφής και επαναπρόθεσης, γιατί η πολιτική γειτονία ε, κατ' ουσίαν τι σημαίνει καταλήγει σε πολιτική επαναπροωθήσεων. Εάν λοιπόν αυτές οι πολιτικές είναι λανθασμένες, δεν έχει καμία σημασία αν είναι πολιτικές ενωσιακές ή ε, πολιτικές μεταξύ κρατών. Παραμένουν αποτυχημένες. Και γιατί είναι αποτυχημένες είναι αποτυχημένες γιατί κατ' ουσίαν τι είναι, είναι πολιτικές νεοαπικιοκρατικές αποφασίζουν δηλαδή κάποιοι να μπλοκάρουν τους ανθρώπους να τους αφήσουν να παραμείνουν εκεί που ζουν μέχρι και να πεθάνουν Υπάρχει κάτι που είπατε ε, κύριε Γκαμπρίτσι ότι αυτοί οι πληθυσμοί θα πρέπει να οριμάσουν. Μα τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι όλοι αυτοί είναι ανώριμοι, είναι παιδάκια. Αυτή είναι μια συμπεριφορά νεοαπικιοκρατική και περνάω τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τη σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η συνθήκη για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δεχτεί, έχει στα χέρια της κάποιες γνωμοδοτήσεις για τη Λιβύη από τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Από τον προηγούμενο Δεκέμβρη όλα αυτά αγνοήθηκαν συστηματικά και χαράσουμε μια πολιτική ενάντια σε αυτά που μας συμβουλεύουν οι διεθνείς οργανισμοί. Δίδουμε κάποια χρήματα για να αναχαιτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους για να τους αναγκάσουμε να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί στις φυλακές της Αφρικής. Έτσι εγώ με λίγα λόγια θέλω να πω η Ιταλία τα ξέρει όλα αυτά, τα γνωρίζει. Αυτή ακριβώς ε, είναι η πολιτική που ακολουθούσε η φασιστική Ιταλία όταν ε, δεν γνώριζε κατ' ουσίαν τι ακριβώς επιδιώκει η Λέγκα του Βορρά. Ευχαριστούμε κύριε Βαλέρο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ έχω πολλές ερωτήσεις για τον κύριο Καμπρίτσι, αλλά οι άλλες ομιλήτριες ουσιαστικά τις έφεραν στην επιφάνεια. Και γι' αυτό θα αναφερθώ σε αυτά που είπαν. Ναι, πράγματι το πρόβλημά μας είναι ότι χώρες μέλη δεν υποδέχονται πρόσφυγες. Δεν το κάνουμε. Αυτό το πρόβλημα. Είπατε ένα στους πέντε είναι πρόσφυγες στην Ιορδανία και στο Λίβανο ακόμα περισσότεροι νομίζω. Στην Ευρώπη πολύ λιγότεροι. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Δεν επιδεικνύουμε αλληλεγγύη ούτε μεταξύ μας, ούτε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης αναφερθήκατε σε μια ε, συνολική αλλά κάρτα λύση. Στην πράξη είναι αλλιώς τα λόγια και αλλιώς την πράξη. Πολλές φορές ακούμε ωραία λόγια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά βλέπουμε στην πράξη όλα αυτά που είπαν οι δύο ομιλήτριες, ότι τελικά κάνουμε τα πάντα για να κρατήσουμε τον κόσμο αυτόν έξω από τις χώρες μας. Αυτό μας ενδιαφέρει λοιπόν, να βρούμε νόμιμες οδούς να φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ανθρωπή. Κυρία Ποντό στους νόμιμους τρόπους. Και αυτό αφορά όχι μόνο τους ανθρώπους που φεύγουν από τον πόλεμο, αλλά που φεύγουν και για άλλους λόγους, για να βρουν δουλειά. Πολλοί άνθρωποι έρχονται και ακούσαμε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τις δικές τους οικονομίες αυτό, ε, τα εμβάσματα που στέλνουν και αυτοί είναι άνθρωποι χωρίς υψηλά προσόντα. Συνεπώς πρέπει να βρούμε τρόπους νόμιμους για να έρχονται εδώ και άνθρωποι υψηλών προσόντων που θέλουν να μεταναστεύσουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να επιδείξουμε περισσότερη αλληλεγγύη και μεταξύ μας και απέναντι σε αυτούς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μαρή Κριστίν Βεριά τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τους ομιλητές. Πολλά υπόθηκαν. Εγώ θα ξεκινήσω από κάτι με το οποίο συμφωνώ και νομίζω ότι όλοι πρέπει να προσέχουν όταν μιλάνε για αυτά τα ζητήματα. Είπατε ότι πρόκειται για κάτι τελικά αρνητικό που κάνουμε. Τα νούμερα αυτό δείχνουν. Τον έχουμε ολιστική, συνολική προσέγγιση επίσης είναι σωστό πρέπει να γνωρίζουμε την πραγματικότητα του συνόλου, επιμένω σε αυτό, του συνόλου της μετανάστευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην επικεντρωνόμαστε ακόμα και στον τίτλο της σημερινή ακρόασης, επικεντρωνόμαστε μόνο στην παράτυπη μετανάστευση όταν μιλάμε για μετανάστευση. Όσο βλέπουμε έτσι τα πράγματα, τότε θα χρησιμοποιούμε λάθος γλώσσα. Γιατί μετανάστευση μιλάμε σήμερα. Μιλάμε για την παράτυπη, μιλάμε για αυτή που μας έρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες, ε, για τη μετανάστευση που μας φτάνει όταν δεν υπάρχουν νόμιμοι οδοί μετανάστευσης. Μα είναι πολύ βασικό αυτό. Αν λοιπόν έχουμε μια συνολική προσέγγιση, αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Μετανάστευση, όταν κάνουμε τον απολογισμό, το είδαμε και χθε είναι θλιβερό. Γιατί το 2015 υπήρχαν τέσσερις λύσεις και το είπατε κι εσείς. Όταν βλέπουμε πώς προχωρούν τα πράγματα, προχωρούν μόνο στην πτυχή της καταστολής, στον έλεγχο των συνόρων, στις επιστροφές. Εντάξει, ωραία, τα λέω λίγο κι εγώ όπως τα είπατε κι εσείς σαν καρικατούρα, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Και πιστεύω πράγματι πως όσο δεν έχουμε αυτή την ισορροπία θα συνεχίσουμε να επιτρέπουμε στους λαθροδιακινητές να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητη και να βρίσκουν νέους δρόμους. Χτες διάβαζα ότι τώρα από την Τουρκία πάνε στην Ιταλία με γιότ, με ιστιοφόρα, με 6.000 το κεφάλι. 6.000 πρέπει να πληρώσει κανείς για να το κάνει αυτό. Όσοι έχουν τα λεφτά λοιπόν. Και οι άλλοι πάνε από την Αλγερία στη Σαρδινία και χωρίς να μιλήσουμε για την έρημο βέβαια, η οποία αποδεικνύεται όλο και πιο επικίνδυνη και θα μας κάσει στα μούτρα και τότε τι θα πούμε όταν έχουμε όλο και περισσότερες εκθέσεις που μας λένε ότι στη Σαχάρα πεθαίνουν περισσότεροι άνθρωποι από όσοι πνίγηκαν στη Μεσόγειο. Τι θα κάνουμε, πώς θα αντιδράσουμε, τι θα πούμε τότε, τι θα κάνουμε, τις πολιτικές μας θα τις μεταφέρουμε ακόμα πιο νότια. Δεν γίνεται. Ερωτήσεις τώρα. Όντως θέλω να μου μιλήσετε για τη Λιβύη και για την πολιτική απέναντι στην Λιβύη. Εγώ ήμουνα στην Τινησία το Σεπτέμβριο με τον Πρόεδρό μας και είδαμε ποια είναι η πραγματικότητα των πολιτικών μας εκεί. Δεν δουλεύουν, μας το είπαν ξεκάθαρα. Μόνο μετατοπίζονται οι διαδρομές, τίποτα άλλο. Επίσης θέλω να ξέρω οι πολιτικές αυτές πώς θα ενηλικιωθούν, πώς θα γίνουν πραγματικές πολιτικές συνεργασίες πώς θα ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού και πώς μπορούμε να έχουμε ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες στα πλαίσια αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού όσο οι δικές μας χώρες μέλη θα συνεχίζουν να έχουν προνομιακές ε, σχέσεις με, για να το πω έτσι γρήγορα, δικτάτορες. Δείτε τι έγινε και στην Καμπόν. Λοιπόν, η μόνη λύση είναι αυτά που ανέπτυξαν οι δύο μιλήτρες, να έχουμε μια πραγματική πολιτική μετακίνησης του πληθυσμού. Και αυτό ετοιμάζοντας τη Διεθνή Συμφωνία για την Μετανάστευση να φροντίσουμε να έχουμε ένα πραγματικό δικαίωμα στη μετακίνηση. Αλλιώς δεν θα καταλήξουμε σε τίποτα. Αν το άρθρο τη Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρεται σε αυτά τα ζητήματα, είναι ακριβώ γι' αυτό. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο να έχουν το ίδιο δικαίωμα να μετακινούνται. Και αν θέλουμε να τηρούμε τις αξίες μας, πρέπει να συμμορφωθούμε προς αυτό ακριβώς το άρθρο και εμείς οι Ευρωπαίοι. Ευχαριστούμε. Ποιο άλλος? Δεν είχα πλήρη κατάλογο ομιλητών. Ωραία. Μάλιν Πιόρκ. Πριν από την κυρία Ενστάιν. Ωραία. Μάλιν Πιόρκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ επίσης ε, και τους ε, δύο προσκεκλημένους ομιλητές ή μάλλον τους όλους προσκεκλημένους ομιλητές. Θέλω να πω ότι ε, με βάση αυτά που άκουσα από την εκπρόσωπο της Κάριτας και του της κυρίας Λάξ ε, αυτή η ιδέα της ε, εταιρική σχέσης ε, αυτό κατ' ουσίαν αυτή η λέξη δεν σημαίνει τίποτα δεν είναι ακριβώς αυτό που θα θέλαμε όλοι μας να βιώσουμε ως εταιρική σχέση ή ως μορφή συνεργασίας βλέπουμε ότι σε αυτή τη συνεργασία κυριαρχεί, κυριαρχεί το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσης, οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ περιορισμένες, αφορούν μόνο ε, τις ε, μεταναστευτικές ροές και αυτά δεν είναι ιδιαίτερα θετικά. Επίσης, για μένα είναι σοκαριστικό το να ακούμε ότι πρέπει να οριμάσουν οι ε, λαοί της Αφρικής και γι' αυτό αντέδρασε και η παρακαθήμενη μου για μένα αυτό είναι νεοαπικιοκρατική γλώσσα, το να πιστεύουμε δηλαδή ότι, μάλλον να το πω αλλιώ, εμείς είμαστε εκείνοι που χαράξαμε τα σύνορα παλαιότερα στην Αφρική. Τώρα τα κάνουμε, θα ξαναπάμε και θα χαράξουμε νέα σύνορα. Ε, πρέπει να συλλογιστούμε λιγάκι, να ανατρέξουμε στην ιστορία μας και να καταλήξουμε στο ε, τι πρέπει να συμβαίνει. Ε, γιατί ε, αυτή τη στιγμή ε, τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα θετικά και νομίζω ότι πρέπει να επανέλθουμε και σε θέματα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου στη σχέση μας με αυτές τις χώρες. Νομίζω σήμερα δεν έχουμε καταλήξει αυτό. Η Σοφή είπε ότι θα πρέπει να δούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι ακριβώς κάνουμε. Να δούμε κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και θα πρέπει επίσης και να σταματήσουμε, γιατί όχι, τη χρηματοδότηση του καταπιστευματικού τεμείου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής, αλλά και την στρατιωτικοποίηση. Και αυτή να την καλέσουμε, γιατί και αυτό εντάσσεται στη συμφωνία που έχουμε συνάψει. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πολλή δουλειά και σοβαρή δουλειά να κάνουμε και πρέπει να την ξεκινήσουμε μετά τη ε, σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που ακούσαμε. Συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά που αναφέρθηκαν από την κυρία Μορένο Λάξ και από την κυρία Μποντό. Το 86% όλων των εκτοπισμένων φιλοξενούνται σε αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει ευθύνη της Ιταλίας για το τι συμβαίνει. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, έχει στείλει μία επιστολή στην ε, κυβέρνηση Ιταλίας υπενθυμίζοντας την απόφαση Χίρση τον Νοέμβρη. Πέντε μετανάστες ε, έχασαν τη ζωή τους και ένα παιδάκι ε, διότι ε, στις λιβικές ακτές παρεμποδίστηκε η Sea Watch να διασώσει τους ανθρώπους αυτούς. Επίσης και χθες κάποια κάποιοι προσπάθησαν να παρέμβουν για να διασώσουν ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα, αλλά χρειάστηκαν τέσσερις ώρες για να μπορέσουν να πείσουν τη Λιβική εκτοφυλακή να του αφήσει να επέμβουν. Όσον αφορά ε, το πλαίσιο, το μεταναστευτικό, το MPF, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, νομίζω ότι παραγωνίζεται πλήρως. Αυτό που βλέπουμε είναι το εξής ότι όλες οι πολιτικές της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορούν ακριβώς την εξωτερική διάσταση, το να αναθεωρείται το θέμα των μισθών κάτι που είναι έξω από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ε, ε, η Κομισιόν τελικά προτείνει αυτούς τους ελέγχους ε, μία αποδοχής, κατά την άποψή μου αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Εγώ προείσταμαι τις ομάδες εργασίας ε, για θέματα μετανάστευση τη επιτροπή ανάπτυξη. Επιτροπής Ανάπτυξης και εμείς έχουμε εκφράσει ανησυχίε μα σε δύο θέματα τα οποία τα αναφέρατε. Ε, οι προποθέσει για τη διαχείριση των συνόρων είναι απαράδεκτες, επικίνδυνες, ε, ε, και αντιβαίνουν στο άρθρο 108 της συνθήκης όπου αναφέρεται ότι ο βασικός στόχος είναι η εξάλληψη της φτώχειας. Όμως ε, όσον αφορά τη Λιβύη και τον Ιγύρα προφανώς εμείς αυτά που κάνουμε δεν στοχεύουν στο να εξάλληψουν τη φτώχεια αλλά στο να διχειριζόμαστε τα σύνορα και να δημιουργήσουμε ε, κάποιες δυνατότητες προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα δηλαδή τα χρήματα κατευθύνονται προς τον έλεγχο των σύνορων και αυτό δεν είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο κάνουμε. Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι ότι μέσα από αυτή την προσέγγιση ε, κινδυνεύουμε να ε, ε, είναι επικίνδυνο κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στη θέση μας με, τους, με τις χώρες Αφρικής και από την άλλη ε, έχουμε σχέσεις ε, με χώρες οι οποίες έχουν μεταναστευτικές ροές ε, προς την Ευρώπη. Ξεχνάμε όλες τις άλλες. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι αυτή η προσέγγιση όχι μόνο είναι αποτελεσματική αλλά επιδεινώνει και την κατάσταση διότι προσπαθώντας να αναχαιτήσουμε τη μετανάστευση από την Αφρική με τον ίδιο τρόπο πλητούμε τις αφρικανικές οικονομίες ε, που βασίζονται στην ελεύθερη μετακίνηση. Άρα δηλαδή μακροπρόθεσμα ε, δημιουργούμε χειρότερα προβλήματα και νομίζω ότι πρέπει πάρα αυτά να αναχαιτήσουμε τέτοιου είδους ε, πολιτικές. Η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως αυτά που θα πω θα διαφέρουν λίγο από τους προηγούμενους. Θέλω να ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές, διότι μπορεί να μην συμφωνώ με κάθε έκφραση και ιδέα που εκφράσατε. Αυτό που κατανόησα όμω είναι ότι και οι τρει ομιλητέ εξήγησαν καθαρά ότι μόνο στοχεύοντα στο κλείσιμο των συνόρων μα και μόνο στοχεύοντα σε επιστροφές δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Διότι εδώ και αιώνε η μετανάστευση λαμβάνει χώρα με διαφόρους τρόπους και για διάφορους λόγου και δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Αν προσπαθήσουμε να τη σταματήσουμε κλείνοντα τα δικά μα σύνορα ή προσπαθώντας να τα μεταθέσουμε προς τα έξω, το μόνο που θα γίνει θα είναι να αυξηθεί η τιμή της μετανάστευσης και δεν μιλώ για τα χρήματα που πληρώνουν στους διακινητές, μιλώ ότι θα αυξηθεί, εννοώ ότι θα αυξηθεί και ο κίνδυνος και ότι οι διακινητές θα χρησιμοποιούν ακόμη πιο βία μέσα. Αυτό νομίζω είναι το κοινό συμπέρασμα από τα όσα είπαν και οι τρεις ομιλητές, βέβαια ίσως να μην το μοιράζονται όλες οι χώρες μέλη μιλούμε για επιστροφές και κλείσιμο των συνόρων και χρησιμοποιούν την αναπτυξιακή βοήθεια για να ασκήσουν πίεση. Αυτό που γίνεται όμως είναι ότι χάνουμε τον σεβασμό που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες χώρες. Χάνουμε τον σεβασμό ως μια ήπειρος ισχυρή, αλλά και μια ένωση που βασίζεται σε αρχές δημοκρατία, ελευθερία για όλους τους πολίτες Εάν τελικώς δώσουμε την εντύπωση ότι αυτά ισχύουν μόνο για του Ευρωπαίους πολίτες και ότι δεν υποστηρίζουμε άλλου να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να αποδώσει. Η δημιουργία μια εταιρικής σχέση δεν είναι μονάχα ζήτημα χρημάτων. Και οι τρει τα είπατε αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται να βρεθούν τρόποι να δοθούν οι δυνατότητε νόμιμη μετακίνηση διευκόλυνση για την έκδοση προξενικών θεωρήσεων, νόμιμη δίαπλη και άδειε εργασία. Με παράδειγμα από τη χώρα μου, τη Γερμανία, είναι εκπληκτικό ότι σε αυτές, τις, μέσα σε αυτέ τι καταστάσει, ορισμένοι Ορισμένε επιχειρήσει πηγαίνουν στην Κίνα για να βρουν ανθρώπου που θέλουν να έρθουν να εργαστούν στην Γερμανία. Αντί να ψάξουν να βρουν ανθρώπου που μπορεί να έρθουν από την Αφρική. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ασκήσουμε πίεση στι ίδιε τι χώρε μέλη μα για να συμφωνήσουν με τις απόψεις αυτές και να λάβουν τα αναγκαία βήματα. Τι πρέπει να κάνουμε για να ασκήσουμε πίεση στις χώρες μέλη, ώστε αντί να παραμένουμε στα σταυρωμένα χέρια και να λέμε «Αχ, τι δύσκολο που είναι», να κάνουν κάποια πράγματα, γιατί για να είμαστε έντιμοι, και αυτό είναι προσωπική πολιτική μου θέση, όταν βλέπω ότι όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ δεν κάνουμε τα σωστά αναγκαία βήματα για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση αυτή, νομίζω όλες οι κυβερνήσεις μας, και δεν κάνω απολύτως και μια εξαίρεση, όλες οι κυβερνήσεις μας είναι ανίσχυρες. Δεν είναι ισχυρές κυβερνήσεις. Δεν αντιμετωπίζουν σωστά τις προκλήσεις. Να πούν στους πολίτες, ναι, είναι δύσκολο. Είναι σημαντική πρόκληση. Δεν θα βρούμε βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα μια λύση, αλλά προσπαθούμε. Δώστε μας εμπιστοσύνη, δείξτε μας εμπιστοσύνη, θα βρούμε λύση. Κάνουμε βήματα και θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε την κατάσταση. Δεν το κάνουν αυτό. Αργούν. Δεν αντιμετωπίζουν την πρόκληση. Χρειαζόμαστε λοιπόν πράγματι περισσότερη Ευρώπη και περισσότερη ανάληψη ευθύνη και στι εξωτερικέ δράσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τι χώρε μέλη. Σα ευχαριστώ. Τέλο, πριν επανέλθουμε στου ομιλητέ μα, η κυρία Μόνμπεργκ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές, ομιλητή και δύο ομιλήτριες καλύτερα, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της κατάστασης. Το πρώτο πράγμα που έρχεται στο νου μου είναι το ζήτημα των επιστροφών, που είναι τόσο σημαντικό και ιδίω μια χώρα όπως η δική μου, η Σουηδία. Έχουμε 18.000 ανθρώπους που θα πρέπει να επιστρέψουν, σημειώνοντας τόσο σημαντικά προβλήματα. Ακούσαμε ήδη στην αίθουσα ότι και εμείς είμαστε ε, αντίθετοι με τις αναγκαστικές επιστροφές, αλλά τι θα κάνουμε αλλιώς όταν έχουμε την κατάσταση αυτή, όταν έχουμε ζητήσει, έχουν ζητήσει οι αρχές από τους ανθρώπους αυτούς να αποχωρήσουν μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Και η Σουηδική νομοθεσία λέει ότι δεν μπορεί να εξαναγκαστεί ο παράτυπος μετανάστης να αποχωρήσει. Χρειαζόμαστε συμφωνία λοιπόν με τις χώρες αυτές για τις επιστροφές. Σκεπτόμουν αυτό που είπατε σχετικά με τα εμβάσματα. Μιλήσατε για κάποιο 13%. Εγώ μάλιστα θεωρώ ότι είναι υψηλότερο, τουλάχιστον για τη Σουηδία. Είδα και ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με οικογένειε στις χώρες αυτές. που στέλνουν το παιδί ξανά και ξανά στην Ευρώπη για να στηρίξει την οικογένεια. Ναι, θέλουν να γίνει αυτό διότι έχουν δει ε, τους γείτονες να το κάνουν. Συνήθως είναι ο γιος της οικογένειας ο οποίος, ε, ο οποίος έρχεται στην Ευρώπη, περιμένει να γίνει δεκτή η αίτησή του. Ε, εν τω μεταξύ η αίτηση ασύλου ενδεχομένω, εν τω μεταξύ δουλεύει παράνομα στην ε, αγορά εργασία, στέλνει χρήματα στην οικογένεια. Μιλάτε πολύ για νόμιμες οδούς μετανάστευσης και εδώ στην παρουσίασα. Νομίζω όμως ότι κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να κρίνει μόνη της αν θέλει να δεχθεί ένα ποσοστό νόμιμων μεταναστών. Θεωρείτε, θεωρείτε όμως ότι η παράνομη μετανάστευση θα σταματήσει μόνο εάν και μόνο επειδή θα δοθούν κάποιες νόμιμες οδοί. Θα εμποδίσουμε τις χιλιάδες μετανάστες να έρχονται στην Ιταλία ή στην Κύπρο. Δεν θα σταματήσει αυτό μόνο και μόνο επειδή θα υπάρχουν νόμιμοι διάβλοι ε, μετανάστευσης. Το έχετε σκεφτεί αυτό. Ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Καπρίτσι στις, για ε, τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τις δύο άλλες ομιλήτριες στα όσα είπαν. Η μόνη όμως παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι όσα είπαν είναι σωστά, αλλά θα πρέπει να ενταχθούν σε κάποιο πλαίσιο, διότι είναι τμήματα μόνο του συνολικού παζλ και δεν είναι το σύνολο. Θα ήθελα, αν με επιτρέπετε, να επιστρέψω σύντομα στη διάσκεψη κορυφή του 99 στο Τάμπερε η πρώτη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφή για θέματα εσωτερικών εσωτερικών δικαιοσύνη κλπ. Τότε και η πρώτη φορά που διορίστηκε επίτροπος ήταν ο Πορτογάλος Βιτορίνο τότε πολλοί από εσά του νέου δεν τον θυμάστε. Εγώ τον θυμούμαι καλά γιατί ήμουν εκπρόσωπό του, εκπρόσωπο τύπου και έγραφα τα ανακοινοθέντα τύπου και στα ανακοινοθέντα τύπου τότε που βγάζαμε 99, ξαναλέω, Ευρωπαϊκό Κοινό Σύστημα Ασύλου. Χρειαζόμαστε γιατί αλλιώ δεν πάμε πουθενά. Δεύτερο, θα πρέπει να γίνει με αλληλεγγύη μεταξύ όρων των χωρών μελών, περιλαμβανομένων και ελέγχων των συνόρων και ούτω καθεξής, για να μπορούν να ελέγχονται όσοι προσέρχονται παράτυπα στα hot spot, αλληλεγγύη, μετανάστες ή πρόσφυγες κλπ. Υπήρχε και ένας άλλος τομέας, πολύ σημαντικός και ενδιαφέρον. Είχαμε πει τότε, εξετάστε τα πραγματικά νούμερα, εξετάστε την πραγματικότητα. Αν βγείτε στους δρόμους και ρωτήσετε σε ένα βελγικό κατάστημα ποιο είναι το ποσοστό ανθρώπων που έρχονται και διαμένουν παράνομα από τη Λιβύη, θα σας πούν 20, 30, 40%. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό. κατά μέσον όρο και θεωρητικό γιατί, γιατί είναι παράτυπη αλλά δεν είναι καθαρά γνωστό. Είναι λιγότερο 5% λοιπόν. Πάντα στο Ζάβεντεμ όπου έρχονται άνθρωποι φτάνουν με παράτυπες ε, βίζες και μετά ξεπερνούν τη διάρκεια της βίζας και ούτω καθεξής. Θα μπορούσα να συνεχίσω να σας λέω σχετικά επιχειρήματα, έχω και ένα άλλο στοιχείο. Οι νόμιμες οδοί. Ξαναέρχομαι στο 1999 στο Τάμπερε. Έγραψα εγώ ίδιος το ανακοινωθέν τύπου και κοιτώζω την κυρία Σλάιν γιατί ήταν και παράξενη κατάσταση τότε στην Ιταλία. Είχε γίνει μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, θεσπιστούν νόμιμες οδοί μετανάστευσης. Γιατί είναι και ζήτημα προσφοράς και ζήτησης ε, εργασίας στην ε, Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Και μία από τις προτάσεις που είχαν γίνει ήταν να γίνει προσπάθεια να έρχονται εποχικοί εργαζόμενοι νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδίω για την Ιταλία, άνθρωποι που θα έρχονταν από την ε, υποσαχάρη Αφρική για την εσωδία τη Στομάτας Πρόταση λοιπόν που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο πρώτη ήταν τότε πρόεδρο, μάλλον αριστερό, και τότε υπήρχε και μια παράξενη σύμπτωση από τι 15 χώρε μέλη, οι 13 είχαν αριστερέ κυβερνήσει και μόνο δύο δεν είχαν. Αυτό είχε συμφωνηθεί τότε από όλε αυτέ τις κυβερνήσει. Και τότε, την στιγμή που πρόκειται να εφαρμοστεί, άλλαξε η κυβέρνηση στην Ιταλία και βγήκε ο Μπερλουσκόνη. Και η αντιπολίτευση στην Ιταλία για να ισχυριστεί ότι ο Μπερλουσκόνη κάνει ανοησίες, το έριξε το νομοθέτημα αυτό. Θα ερχόντουσαν οι άνθρωποι αυτοί, θα δούλευαν τρει-τέσσερι μήνε, θα έβγαζαν αρκετά χρήματα για να ζήσουν τι οικογένειέ του ολόκληρο το χρόνο και οι Ιταλοί αγρότε θα είχαν και την ευκαιρία να πούν έλα ξανά του χρόνου και εδώ και χαιρετισμού στη γυναίκα σου. Τα λέω κάπως ε, με απλό τρόπο, αλλά αυτό είναι ένα πρώτο μήνυμα που έχω να σας πω. Εδώ και 20 σχεδόν χρόνια που είμαι στη δουλειά αυτή και μπορώ να σας πω ότι συμφωνώ μαζί σας σε μια σειρά επιχειρημάτων που προβάλλατε. Το πρόβλημα όμως είναι δεν είναι τα θεσμικά όργανα που δεν κατέθεσαν προτάσεις υπάρχει έλλειμμα ανάληψης ευθύνης από τις χώρες μέλη. Και μπορείτε να το καταλάβετε αυτό, διότι για θέματα που έχουν σχέση με το μεταναστευτικό μπορούν να οδηγήσουν κυβερνήσει να κερδίσουν ή να χάσουν τις εκλογές. και αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σα. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουν σε προτάσεις με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατατεθούν στο τραπέζι και να αναλάβουν ευθύνε οι κυβερνήσει. Και τότε Κάποιος είπε τι μπορούμε να κάνουμε ως ευρωβουλευτές. Ως ευρωβουλευτές, ευρωβουλευτές είσαστε, αλλά είσαστε και επίκοοι των χωρών μελών σας. Νομίζω λοιπόν ότι μπορείτε να πιέσετε και μέσα από τα κόμματά σας, τα εθνικά σας κόμματα, να, να πιέσουν και αυτοί με τη σειρά τους, τις κυβερνήσεις, όταν έρχονται στις Βρυξέλλες, να στηρίξουν, εάν και όταν, θα καταθέσουν κάποια ευφύη πρόταση τα θεσμικά όργανα να την υποστηρίξουν. Το δεύτερο, όταν μιλώ για ολιστική προσέγγιση 360 μοιρών, διότι επικρίθηκα πολύ στις παρεμβάσεις σας, λέτε ότι ρίχνουμε όλο το βάρος στις επιστροφές. Το πρώτο πράγμα που είπα όταν άρχισα την παρέμβασή μου ήταν το μήνυμά μου δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσει κανείς θέματα μετανάστευσης, κινητικότητας, μετακίνηση πληθυσμών χωρίς μια σοβαρή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Και πέραν της μετανάστευσης συμφωνώ μαζί σας όταν λέτε στο ευρωπαϊκό έγγραφο που αδιαβάσατε λέει ότι ναι, ναι, κυρίως βάζετε στις επιστροφές. Μα αυτά τα λένε ορισμένα υπουργεία των εξωτερικών. Αν διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο θα δείτε κάπου αλλού να λέει, εμείς ήμασταν αυτοί, Μογκερίνη δηλαδή, ωραία όλα αυτά αν θέλετε, διότι χωρισμένοι είσαστε και θέλετε να κάνετε επιστροφές, αλλά θα πρέπει να τις εντάξετε σε μια ε, διμερή ατζέντα, διμερές θεματολόγιο εξωτερικών σχέσεων. Θα πρέπει να εξετάσετε λοιπόν τι λένε τα θεσμικά όργανα και πάντοτε υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι εν τέλει οι χωρισμένοι είναι αυτές οι οποίες συμφωνούν και θα δούμε σε ποιο βαθμό μπορούν να συμφωνήσουν στις προτάσεις των θεσμικών οργάνων. Και αυτό βεβαίως που θα αποφασίσουν πρέπει και να στηριχθεί και να τροφοδοτηθεί. Διότι απλώς άσκηση κριτικής, καλώς, σύμφωνη και εγώ συμφωνώ με την κριτική σας, αλλά πρέπει να βρούμε και τρόπο να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν ε, αυτές οι άλλες παρατηρήσεις που έγιναν για τη μετανάστευση κατά αν αυτή θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εξωτερικής πολιτικής θα μου επιτρέψει εδώ να ανοίξω μια παρένθεση και να αναφέρω μια πολύ συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρθηκα σε αυτήν όταν είπα ότι χάσαμε το τρένο μετά την 11 ε, Σεπτεμβρίου 2003 η κρίση πατέρα Μαρόκο-Ισπανίας θα θυμάστε όλοι σας ε, είναι περίπου και σήμερα το ίδιο που συμβαίνει αλλά σε μικρότερη κλίμακα πραγματικά άνθρωποι πέθαναν στι ακτέ και τότε η Ισπανία δεν μπορούσε να λύσει το πρόβλημα σε διμερέ επίπεδο με το Μαρόκο. Και η Ισπανία ζήτησε από τα άλλα κράτη-μέλη να αναθέσουν στην Ισπανία τη δυνατότητα τη επαναπρόθεση. Αυτή λοιπόν είναι η περίφημη προσέγγιση των επιστροφών, το θέμα τη ασφάλεια. Ξεκινήσαμε λοιπόν τι διαπραγματεύσει με του Μαροκινού, πήγαμε να του δούμε και το πρώτο που μα είπαν οι Μαροκινοί είναι ότι συγγνώμη αυτό δεν είναι δικό μα πρόβλημα, δικό σα είναι το πρόβλημα και εν περιπτώσει με τα εμβάσματα των ανθρώπων μας από την Ευρώπη έχουμε περισσότερα χρήματα από αυτά τα λίγα που μας δίνετε εσείς εν είδη αναπτυξιακής πολιτικής και βοήθειας. Μας είπαν βέβαια ότι αν πραγματικά θέλετε εταιρική σχέση, αν πραγματικά θέλετε business, ας προσπαθήσουμε να περάσουμε σε αυτό και ξέρετε τι πρότειναν. Πρώτον, σας παρακαλούμε ε, μη βάλτε διαπραγματεύσεις ε, στους επιχαίους τίτλους ε, των εφημερίδων γιατί μας φαίνεται σε δύσκολη θέση με όλες τις άλλες χώρες Αφρικής. Και μετά είπαν ανεξάρτητα από την Ευρώπη και ανεξάρτητα από τη μετανάστευση εμείς αυτό που χρειαζόμαστε στο Μαρόκο τότε και μετά από αίτημα του Βασιλιά ήταν να επιταχυντούν οι μεταρρυθμίσεις και της κατάστασης κυρίως των γυναικών. Ε, να μεταρρυθμιστεί ο εκπαιδευτικό τομέας, μεταρρυθμιστεί σε θέματα τουρισμού, μεταφορών, ενέργειας, οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν χρειαστήκαμε τρία χρόνια να διαπραγματευτούμε με τους Μαροκινούς για όλες, με όλες αυτές τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξετάσαμε σε όλα τα επίπεδα αυτά που ζήτησαν οι ίδιοι Μαροκινοί, το δικό τους το αναψυακτικό μοντέλο για να προχωρήσουν για να είναι πιο σταθερή και προσπαθήσαμε να δούμε τι μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για προσθέμενη αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι σε διμερές επίπεδο. Φτιάξαμε λοιπόν μία δέσμη και είπαμε Open Sky, συμφωνία. Δηλαδή Ryanair, German Wings και άλλες εταιρείε χαμηλού κόστους θα μπορούσαν να πετάνε στο Μαρόκο. Περισσότερες επενδύσεις στον τουρισμό και πάρα πολλά άλλα. Σε αυτό λοιπόν το πακέτο είχαμε και μία συμφωνία για την Αλία, για τη Γεωργία. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι η εξωτερική διάσταση των κοινοτικών πολιτικών. Η Συμφωνία Open Sky των Ανοιχτών Ουρανών είναι μια συμφωνία νησιακή και ε, αν κάνεις κανείς μια συμφωνία με τρίτη χώρα, αυτό είναι εξωτερική διάσταση. Αυτό αξίζει πάρα πολλά χρήματα, φέρνει πάρα πολλές δουλειές, είναι μια κατάσταση που ωφελεί και τις δύο πλευρές και φέρνει επενδύσεις σε αυτές τις χώρες, φέρνει θέσεις απασχόληση σε αυτές τις χώρες. Κανένα κράτος μέλος ε, ε, δεν ε, μπορεί να το οικειοποιηθεί γιατί είναι μια ευρωπαϊκή συμφωνία. Με λίγα λόγια λοιπόν εμείς ειλικρινά χρειαστήκαμε πολύ χρόνο για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πακέτο που δεν είχε άμεση σχέση με τη μετανάστευση. Είχε ξεκινήσει μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους να μπορεί να εφαρμόσει πολιτική επαναπροωθήσεων ακριβώς και μόνο για την υπόθεση πατέρας. Όμως εμείς αυτή την ευκαιρία την εκμεταλλευτήκαμε. Εκμεταλλευτήκαμε την εντολή των 28 για να μπορέσουμε να ε, έχουμε την εξωτερική διάσταση της ε, ενωσιακής πολιτικής. Για πρώτη φορά λοιπόν προτείναμε στα κράτη-μέλη να χαράξουν μια ε, εξωτερική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό λοιπόν που συνέβη και δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί αν το κάνω θα με απολύσουν αύριο το πρωί αλλά de facto αυτό που συνέβη ήταν το εξή. Οι Μαροκινοί και οι Ισπανοί κατέληξαν σε μια διμερή συμφωνία μια συμφωνία που το Μαρόκο είπε ότι εγώ θα τα ξεκαθαρίσω όλα, δεν θα έχετε πια σχεδίες αλλά και εσείς ε, θα ξεμπλοκάρετε το πακέτο που έχει μπλοκαριστεί στις Βρυξέλλες, Συμφωνία Ανοιχτών Ουρανών και όλα τα άλλα. Ουσιαστικά μας ζήτησαν να ξεμπλοκάρουμε και τη Συμφωνία Ελίας είναι σαφές αυτό γιατί, γιατί οι Ισπανοί ήθελαν να ψαρεύουν στο Μαρόκο. Μόλις λοιπόν ε, τους δώσαμε την ε, Συμφωνία Ελίας, μετά από τρία λεπτά ήρθαν η Ryanair, η German Wings και όλοι οι άλλοι και μα είπαν, ξέρετε κάτι, εμείς δεν είμαστε και βλάκες, θέλουμε και εμείς αυτή τη συμφωνία και άλλη συμφωνία και παράλληλη. Και έτσι λοιπόν ε, κανιβαλίσαμε ειλικρινά την εξωτερική διάσταση της ενωσιακής πολιτικής κανιβαλίσαμε πραγματικά την προσθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα αυτά έγιναν όχι γιατί ο Θαπατέρο ήταν κακός άνθρωπος. Ο Θαπατέρο είχε και τη δική του την εσωτερική πίεση στη δική του χώρα και ήθελε να προχωρήσει γρήγορα. Τα 27 άλλα κράτη-μέλη σας ερωτώ, είναι πραγματικά υπεύθυνα και σήμερα μετά από 15 χρόνια αν είχαμε μια συμφωνία επαναπρόθεσης με το Μαρόκο ως αντάλλαγμα μιας εταιρική σχέσης που συνδέει το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο του Μαρόκου στην ευρωπαϊκή κοινή αγορά δεν θα ήταν καλύτερα να είχαν γίνει όλα αυτά τότε και όχι σήμερα. Η απάντηση προφανώς είναι ναι και γι' αυτό λοιπόν είπα στην παρέμβασή μου ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που περνάει το τρένο και ίσως μπορούμε αυτή τη φορά να το πάρουμε και να μην κανιβαλίσουμε την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνο του. Μόνο ε, ένα κράτος να βρει επαναπρόθεση ή νομικούς ε, διάβλους ε, δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνο στα κράτη-μέλη. Χρειάζονται πακέτο. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Uh, yeah, nothing uh, much is left to say, but um, I would like to Ευχαριστώ και εγώ. Για το θέμα των επιστροφών θα σας απαντήσω. Όπως σωστά είπατε, ακόμα και αν θέλει κανείς να αυξήσει τις επιστροφές, εγώ δεν λέω ότι θα έπρεπε να συμβαίνουν, αλλά λέω ότι αν θα θέλατε να πετύχετε αυτό το στόχο, δεν μπορείτε να το κάνετε μόνο με κοντόφθαλμες συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης. Πρέπει να βάλετε κάτι ουσιαστικό στο τραπέζι πέρα από την μετανάστευση. Ακόμα και οι χώρες που θέλουν να πούνε ότι κοιτάξτε θα αυξηθούν οι επιστροφές, να το ξέρει ο κόσμος, αυτό δεν πρόκειται να προχωρήσει ήπια. Υπάρχει τεράστια υποκρισία σε πολλές χώρες μέλη. Κυρίως στην Νότια Ευρώπη, ε, πολλές ε, χώρες εξαρτώνται από τους μετανάστες που έρχονται και δουλεύουν και τους εκμεταλλεύονται πολύ συχνά και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν θέλετε να έχετε ε, νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να ρυθμίσετε και αυτούς τους τομείς που χρησιμοποιούν οι μετανάστες. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το ότι οι χώρες προσπαθούν μόνες τους να κάνουν πράγματα και μετά έρχεται η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που δίνει κάποια κατεύθυνση και δημιουργείται ένα βραχικύκλωμα. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν μια αντιμετώπιση πιο σφαιρική από αυτήν που κάνει ο κάθε υπουργό Μετανάστευση τη κάθε χώρα χωριστά. Ευχαριστώ. Κύριε Μωρένο Λάξη. Έχω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις να κάνω. Με ρωτήσατε ε, πού οφείλεται η επιτυχία της εξωτερικής δράσης μείωση των ροών δεν θα πρέπει να αποτελεί το μόνο δίκτυ. Πουθενά στη συνθήκη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που υπάρχει είναι τα άρθρα 2 και 21 της συνθήκης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικεντρώνεται στην ποιότητα της μετανάστευσης που λέει ότι θα πρέπει να τυχαίνει η διαχείριση ανάλογα και βάση των δικών μας ιδρυτικών αρχών. Και για να απαντήσω στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τι παρατηρήσει του κ. Καμπριέτη, θα έλεγα ότι καταλαβαίνω, κατανοώ τη θέση τους βεβαίω. και καταλαβαίνω ότι οι στόχοι και η κατεύθυνση των εξωτερικών σχέσεων βέβαια εξαρτάται από τις χώρες μέλη και το Συμβούλιο. Παρόλα αυτά όμως θα έπρεπε να βγούμε από τη λογική των διεθνών σχέσεων που περιορίζονται σε σχέσεις κρατών. Γιατί έτσι υπονομεύεται η θέση των ίδιων των μεταναστών. Και έτσι όπως έχει το διεθνές δίκαιο, ε, υπόκειται με δικαιώματα στο δίκαιο οι μετανάστες. Μπορούν να φύγουν από μια χώρα εφόσον θέλουν, όπως και οποιοδήποτε άλλος. Αν αυτό συνδυαστεί με την αρχή του non-refoulement, σημαίνει ότι πρέπει να έχει δίκαια μεταχείριση οποιοδήποτε, ανεξαρτήτως καθεστώτος το οποίο εμπίπτει. Και για αυτούς που χρειάζονται διεθνή προστασία επιπλέον έχουν το δικαίωμα στο άσυλο. Η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο άρθρο 18 το αναγνωρίζει αυτό. Ξεκάθαρα. Οπότε δεν τίθεται θέμα εδώ πέρα πλαισίου μεταναστευτική συνεργασία ή οτιδήποτε άλλο του Συμβουλίου ή των χωρών μελών που μπορεί να το παρακάμψει αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση από μόνη τη δεν μπορεί αυτό να το παραβλέψει. Οπότε στην ερώτηση τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η χρηματοδότηση, ο έλεγχος των δράσεων όχι μόνο από τις χώρες μέλη, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών, της Frontex για παράδειγμα. Χρήση των συνομοθετικών τους αρμοδιοτήτων για αρχές και θεμελιώδη δικαιώματα προκειμένου αυτά να ξαναμπούν στην εικόνα. Τώρα μάλιστα με το τρίτο πακέτο για το άσυλο που συζητιέται υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μάλιστα σε σχέση και με νέα μέσα διαχείρισης συνόρων, θεωρήσεις κλπ. Και θα καλούσα τους ευρωβουλευτές να αναλάβουν ηγετικό ρόλο που δεν έχουν ε, δεχτεί ούτε χώρες, ούτε το Συμβούλιο, ούτε Επιτροπή, ώστε να μπούμε στο mode κρίση και να φροντίσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Πώς θα πιέζαμε τις χώρες μέλη. Naming and shaming. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Το link που ήθελα να σας δείξω σε βίντεο ακριβώς αυτό κάνει. Να μην τα μόνο με τους εταίρους μας, αλλά και με τις χώρες μέλη. Και ακριβώς με τον χώρο μεταξύ των δύο, η Μεσόγειος να στηρίξουμε ό,τι προσπάθειες γίνονται, στρατηγικές κλπ. Από τον Νοέμβριο του 2017 υπάρχει μια δράση κατά της ε, Ιταλίας για καταχρήσεις που έγιναν στο καταπίστευμα για την ε, Αφρική. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Επίσης να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός ε, διασταυρώσεων ελέγχων για να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε και οι άλλοι και να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαδικασίες επιπαραβάση κάθε φορά που χρειάζεται. Υπήρξε μια ε, προφορική ερώτηση του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή για ένα newsletter της Association Press όσον αφορά τη συνεργασία της Λιβύης με την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι 46 εκατομμύρια δόθηκαν προς την Λιβύη και ότι το Ιταλικό Υπουργείο Εσωτερικών ελέγχει τι γίνεται με τα χρήματα αυτά. Νομίζω εδώ πέρα ότι ο καθένας μπορεί να δει και να διαπιστώσει ότι αυτό δεν είναι αμερόληπτο αν είναι Ιταλοί αυτοί οι οποίοι κρίνουν πώς χρησιμοποιεί τα χρήματα η Λιβύη. Συνεπώ οι ευρωβουλευτέ δεν θα έπρεπε να μένουν ικανοποιημένοι με τέτοιου είδου ε, λύσει και να πιέζουν την Επιτροπή που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων με τη σειρά τη να πιέζει και να ελέγχει οι καταστάσει. Τέλο, αν οι νόμιμε δύο διμετανάστευση θα σταματούσαν την παράνομη μετανάστευση. Αυτά που είπε η Σουδέζα συνάδελφο. Σε αντίθεση με αυτό που εκείνη λέει, η εισδοχή δεν είναι κάτι που αποφασίζουν ελεύθερα οι χώρε μέλη. Ήδη το 1987 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι ο έλεγχο εισόδων πρέπει να υπόκειται στι διεθνεί υποχρεώσει, δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα μεταναστών να αποχωρούν, non refoulement και άσυλο. Συνεπώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να φροντίζει να συμμορφώνεται προ του δικού τη νόμου πρώτα απ' όλα και προ το άρθρο 2 τη συνθήκη που, μιλάει, που μιλάει για το σεβασμό της Χάρτας Θεμελιωμένων Δικαιωμάτων. Το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες μέλη το κάνουν όταν εφαρμόζουν ευρωπαϊκό δίκαιο. Υπάρχει προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να αλλάξουμε κατεύθυνση και για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται το πλαίσιο μεταναστευτικής συνεργασίας και για, την, ε, και για όλα τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο μας. Θα έπρεπε να είχατε χρησιμοποιήσει τα 17 λεπτά που σας παραχώρησα. Μπορείτε να απαντήσετε αν θέλετε. Ναι, 30 δευτερόλεπτα για κάποιους που με κατηχώρησαν επειδή είπα out of context πρέσβης σημαντικής αφρικανικής χώρας στη Βαλέτα είπε στις άλλες αφρικανικές χώρες εντός εισαγωγικών θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε όταν θα γίνουμε, όταν θα ενηλικιωθούμε ως κυβερνήσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια νοοτροπία στις ίδιες τις τρίτες αυτές χώρες. Γι' αυτό είναι μια φράση που χρησιμοποίησε Αφρικανός πρέσβης και είπε ότι όταν θα ενηλικιωθούν οι κυβερνήσεις μας θα αποφασίσουμε κτλ. Τα, τα λέω αυτά για να σας φύγει η ιδέα ότι είμαι νέο απεικιοκράτης. Η επικοινωνία είναι το παν, λέει ο Πρόεδρος. Το Τάμπερε ήταν από τα καλύτερα συμβούλια για εσωτερικά και, και ε, δικαιοσύνη και ο Βιτορίνο ήταν από τους καλύτερους επιτρόπους. Δεν νομίζω ότι είχε χρησιμοποιήσει ε, τέτοια φράση ή κανένας από τους ανθρώπους του. Μου φάνηκε πολύ χρήσιμη η συζήτηση και εσείς και η κυρία Μορένο απαντήσατε σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τα προνόμια, με τις εξουσίες του Κοινοβουλίου που έθεσε η κυρία Ιντφέλτ. Έχουμε θέμα με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και το γεγονό ότι παρακονίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συνεχίσουμε να το θέτουμε και να πιέζουμε τι χώρε μέλη. Αυτό είναι άλλωστε ο ρόλο μα του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Άλλωστε προσκαλούμε, καλούμε ξανά και ξανά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων και αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε για να προσεγγίσουμε όλο και περισσότερο ως Επιτροπή ε, Θεμελιωδών Ελευθεριών και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε πέρα του σεβασμού των προνομίων μας όλο και περισσότερο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε όμως τώρα να ακούσουμε τους άλλους προσκεκλημένους. Ήθελα να τα προσθέσω αυτά τα τελευταία λόγια διότι μου φαίνεται ότι είναι κρίσιμα και σωστά είπατε Τερέζα. Να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο πάνελ για τις συμφωνίες κινητικότητας. Αφού πρώτα ευχαριστήσω ωστόσο τους τρεις προσκεκλημένους που αποχωρούν. Θα αλλάξουμε πάνελ και θα σας συστήσω τα πρόσωπα αυτά όταν θα προσέλθουν. Έχουμε την ευκαιρία τώρα να, παρακολου... να ε, ρίξουμε μια, μια κοντινότερη ματιά στις συμφωνίες κινητικότητας. Θα έχουμε τώρα πρώτα τον εξοχότατο Ταχάρ Σερίφ πρέσβη της Δημοκρατίας της Τινησίας στις Βρυξέλλες. Σε ευχαριστώ ε, συνάδελφοι. Έχουμε όπως είπα καθυστερήσει λίγο ήδη αν ο κύριος Πρέσβης είναι έτοιμος να αρχίσουμε πρώτα ακούγοντας τον κύριο Ταχάρ Σερίφ πρέσβη της Δημοκρατίας της Τινησίας της Βρυξέλλες όπως είπε η κυρία Βεργιά προηγουμένως επισκεφθήκαμε πρόσφατα την Τινησία σε μια πραγματικά πολύ ειλικρινή και ανοιχτή αποστολή στην Τινησία χρήσιμη επίσκεψη για να κατανοήσουμε ποιες είναι οι πιέσεις που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή και ποιε είναι οι σχέσεις και με την Λιβύη. Ήταν πραγματικά αποκαλυπτική η αποστολή αυτή. Είδαμε βέβαια και την ακτοφυλακή και, και, και παρακολουθήσαμε και άλλες σημαντικές δράσεις. Σας ευχαριστούμε που είστε παρόν σήμερα εδώ και είναι πράγματι πολύ σημαντικό το θέμα σας. Ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πολύ όλους. Πολύ χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε για αυτήν την συνεργασία για την κινητικότητα και τη διευκόλυνση θεωρήσεων. Το 2014 υπέγραψε και η, την Ισία δήλωση για αυτήν την εταιρική σχέση, η οποία δεν είναι δεσμευτική όμως, γιατί σήμερα έχουμε το δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων για αυτήν την συνεργασία για την κινητικότητα και ανεβλήθη για αύριο αυτή η συνάντηση. Οπότε θα είχα πολύ περισσότερα να σας πω αύριο. Τώρα από πλευράς της αποτελεί άνισμα ανάπτυξης οικονομικής, πολιτιστικής, ενισχύοντας την ανθρώπινη διάσταση εκατέρωθεν της Μεσογείου. Γνωρίζετε ότι σήμερα διαπραγματευόμαστε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ανάμεσα στην Τινησία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια παράλληλη διαδικασία με την κινητικότητα, δηλαδή αυτή των ελεύθερων συναλλαγών και αυτό είναι ενδιαφέρον. Υπάρχουν όμως πολλές ανησυχίες από πλευράς της Τινησίας. Και τι εννοώ. Θα ανοιχτούμε προς ένα γίγαντα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τινησία όμως είναι και αυτή 11-12 εκατομμύρια. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τη γεωργία και τις υπηρεσίες. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες, κυρίως για τη γεωργία διότι γενικά μιλώντας πρόκειται για μικρές καλλιεργούμενες επιφάνειες με έναν ή λίγο περισσότερο, πάντων από οικογένειες καλλιεργούνται αυτές οι γέες και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Υπάρχει λοιπόν τεράστια ανησυχία και για τις υπηρεσίες ισχύει το ίδιο, γιατί θα έπρεπε και εκεί να υπάρξει μια προσαρμογή συνολικά για τις υπηρεσίες. Γιατί ένα γραφείο ε, δικηγορικό στην Τινησία αποτελείται από έναν, εδώ από 100. Ε, με μια απλή ταυτότητα κυκλοφορεί κανείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Τινήσιοι πρέπει να ζητήσουν ε, θεώρηση. Και αν δεν την έχουν και πρέπει επιγόντως να μετακινηθούν, δεν μπορούν. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, οι δύο αυτές συμφωνίες πάνε εκ παραλίλου. Γιατί από τη μία ανοίγουμε την αγορά με τις ελεύθερες αλλαγές, από την άλλη μπλοκάρουμε τον κόσμο. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητέ. Πριν αναφερθήκατε στο Ζάβεντεμ κάποια στιγμή, τελευταία υπάρχουν πολλές επαναπροθήσεις, ρεφουλμό. Γιατί, Γιατί δεν έχουν θεώρηση. Η επανάσταση του 2011 ήταν για την ε, ενότητα και την αξιοπρέπεια, συγγνώμη, για την αξιοπρέπεια. Δεν ήταν τόσο για την ελευθερία, ήταν για την αξιοπρέπεια. Πώς θέλετε, ναι, διπλωματούχοι να περιμένουν 7 και περισσότερα χρόνια χωρίς πόρους, χωρίς δουλειές. Αρχίζει ο κόσμος λοιπόν να σκέφτεται «Α, τελικά πριν την Επανάσταση μπορεί να ήταν και καλύτερα» γιατί τότε είχαμε 5 και 6% ανάπτυξη κάθε χρόνο. Τώρα με το ζόρι έχουμε 1% ανάπτυξη και με 1% ανάπτυξη δεν μπορούμε να πληρώσουμε ε, θέσεις απασχόλησης. Έχουμε 15% και παραπάνω ανεργία στην Τινησία, 650.000 ε, άνεργους, εκ των οποίων οι μισοί έχουν πανεπιστημιακά διπλώματα. Αυτό εξηγεί και το τελευταίο κύμα, το μεταναστευτικό προς την Ιταλία Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αλλά αυτό δεν είναι όλη ιστορία. Οι απελπισμένοι νέοι ή που θα πρέπει να πέσουν στη θάλασσα να πνιγούν ή να πάνε να συνεργαστούν με την ε, ΤΑΣ, με το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε εδώ πέρα ε, να τους ε, βοηθήσουμε, να τους σταθούμε δίπλα τους, γιατί αλλιώ είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Αυτά από το 2011. Οπότε, μιλώντα τώρα για την κινητικότητα. Σε αυτή τη συνεργασία πρέπει να δώσουμε λύση και να καθισκάσουμε αυτές τις ανησυχίες. Πώς να δημιουργηθεί ανάπτυξη στη χώρα, κυρίως στις ε, πιο μειονεκτικές περιοχές, που κάναν την επανάσταση. Δυστυχώς δεν έγιναν αρκετά παρόλο που έχει προχωρήσει αρκετά η πολιτική διαδικασία. Οικονομικά μιλώντας, χρειαζόμαστε πολύ βοήθεια. Για τις θεωρήσεις, Βίζα. Η Τινησία θα προσπαθήσει να διευρύνει τις κατηγορίες που μπορούν να επωφεληθούν από μια τέτοια διευκόλυνση και να φροντίσει να μειωθεί το κόστος, ο χρόνος κλπ. Για την επανεισδοχή για μας η αρχή είναι να την απορρίπτουμε για τρίτους, για επικός τρίτων χωρών. Αυτά λίγο πολύ είχα να σας πω. Αλλά για την παράτυπη μετανάστευση, μετά το κύμα του 2011, είχαμε μια καλή συμφωνία με την Ιταλία. Υπήρξαν πολλές ε, επιστροφές που έγιναν με τη θέληση των ε, ανθρώπων προς την, ε, την Ισία. Ε, βοηθηθήκαμε και για να αγοράσουμε κάποιο εξοπλισμό γιατί έγιναν πολλές καταστροφές στην Επανάσταση. Έχουμε βοήθεια και για την ασφάλεια. Δεν φτάνουν όμως όλα αυτά. Και τελευταία είχα μια συνάντηση με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Home και μου είπε ότι για πρώτη φορά είμαστε έτοιμοι να χρηματοδοτήσουμε εξοπλισμό στην την Ισία. Πριν τίποτα. Είναι για πρώτη φορά και είναι μια νέα ιδέα ε, που έχουμε και ελπίζω και την Ισία να μπορέσει να ανταποκριθεί πολύ γρήγορα. Όλα αυτά για να σας πω ότι την Ισία δεσμεύεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταπολεμήσει την ε, παράτυπη μετανάστευση. Εμείς θα προτιμούσαμε μια μεγαλύτερη διευκόλυνση όσον αφορά τις θεωρήσεις. Στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης και ερχόντουσαν πολύ την ίση στην Ευρώπη για μια εβδομάδα, για ταξίδι, χωρίς πρόβλημα. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Σας ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το έχουμε δει και αυτό το θέμα. Η κυρία Βερζιά ε, νομίζω έχει επισημάνει το θέμα της διευκόλυνσης ε, ε, θεωρήσεων και το πώς το αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο. Πάμε στην επόμενη μιλήτρια, στην κυρία Γκρατσιέλα Ρίτσα από τις Διεθνείς Σχέσεις, Γενική Διεύθυνση Home. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστώ επίσης και τον ε, ε, πρέσβη της Τινησίας, πάρα πολύ καλή παρουσία του, του κυρίου Σερίφ. Εκ μέρου της γενική διεύθυνση ε, εσωτερικών Υποθέσεων θα ήθελα να σας παρουσιάσω το θέμα της συνεργασίας για κινητικότητα. Για να είναι σαφές το τι ακριβώς θέλουμε να σας μεταφέρουμε, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει σχέση με το πλαίσιο κινητικότητας το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως. Ας δούμε λιγάκι τι ακριβώς έχει παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια γενικότερη προσέγγιση σχετικά με τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Αυτά ανάγονται στο 2005 και στο 2011. Υπάρχουν τέσσερις ε, πυλώνες ε, επί των οποίων θα έπρεπε να βασίζεται ο διάλογος για τη μετανάστευση με όλες τις τρίτες χώρες συγκεκριμένα νομότυπη μετανάστευση, ε, παρεμπόδιση της παράνομης μετανάστευσης, ε, παροχή ασύλου και μεγιστοποίηση των ε, ε, προεκτάσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Είχαμε λοιπόν το πλαίσιο αυτό συνεργασία, το οποίο κατ' ουσίαν τι είναι, είναι ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται η μετανάστευση, όχι όμως ε, προβάλλοντας ιδιαίτερα τη μετανάστευση, αλλά προβάλλοντας ε, κυρίως ε, άλλες πτυχές. Και αυτό νομίζω ότι παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ομιλία. Όταν λοιπόν εγκρίθηκε αυτή η προσέγγιση για την κινητικότητα, κατ' ουσίαν υπήρχαν δύο εργαλεία, τα οποία τότε είχαμε προγραμματίσει. Το ένα εργαλείο ήταν η συνεργασία για θέματα κινητικότητας και το άλλο ήταν η κοινή ατζέντα για τη μετανάστευση και την κινητικότητα. Ας δούμε ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε αυτά τα δύο εργαλεία. Η συνεργασία κινητικότητας υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη και η συμφωνία αυτή εστιάζει περισσότερο σε ανάληψη ευθυνών. Ενώ η κοινή προσέγγιση για τη μετανάστευση και την κινητικότητα υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ μέρους όλων των κρατών μελών ε, αυτή η συμφωνία έχει υπογραφεί με την Αιθιοπία, την Ινδία και την Ιγυρία. Και συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη Βραζιλία. Θα ήθελα λοιπόν να εστιάσω στην ε, συνεργασία για θέματα κινητικότητας και να έχει την καλοσύνη να πάτε πίσω στην προηγούμενη διαφάνεια για να δούμε λιγάκι τη χρονική εξέλιξη. Αυτή η συμφωνία θα έπρεπε αρχικά να υπογραφεί το 2008. Την επόμενη χρονιά, το 2018, θα οργανώσουμε μία εκδήλωση για να κάνουμε απολογισμό και για να δούμε και τι θα γίνει στο μέλλον. Το 2008 υπογράφηκε συμφωνία με το Πράσινο Ακροτήρι και με τη Μολδαβία. Μέχρι το 2013 ε, αποδόθηκε ιδιαίτερη σημασία κυρίως στις ανατολικές χώρες. Και το 2013 υπογράφηκε η συμφωνία με το Μαρόκο, με το Αζερμπαϊτζάν, το 2014 με την Τινησία και την Ιορδανία και πέρυσι υπογράφηκε η συμφωνία με τη Λευκορωσία. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της ε, συνεργασίας. Στόχος είναι να υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο για διμερή συνεργασία σε θέματα μετανάστευσης και κινητικότητας. Να υπάρχει δηλαδή μια ολιστική προσέγγιση. Γιατί η ολιστική προσέγγιση, γιατί κατ' ουσίαν ε, εξετάζουμε τα αίτια, τα βασικά αίτια της ε, τα χαρακτηριστικά αυτού του πλαισίου είναι ότι δεν είναι νομικά δεσμευτική αυτή η συμφωνία. Ε, η συμφωνία είναι κομμένη και ραμμένη στις ανάγκες των ε, ε, μελών και των χωρών που υπογράφουν τη συμφωνία, γιατί παραδείγματο χάρη η Λευκορωσία έχει τελείω διαφορετικέ ανάγκε από την Τινησία ή το Μαρόκο. Υπάρχει ευελιξία, προσαρμοστικότητα σε αυτή τη συμφωνία και η βασική ιδέα είναι να προκύψει μια κοινή προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Αυτό νομίζω ότι συζητήθηκε εκτενώς ε, στο προηγούμενο κομμάτι της ε, συνεδρίας μας, εκεί όπου έγινε λόγος ε, για την σχέση της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και κρατών μελών. Εμείς, όπως σας είπα, ασχολούμεθα με τους πυλώνες αυτής της συμφωνίας και μας ενδιαφέρει επίσης και η ε, διευκόλυνση στην ε, χορήγηση θεωρήσεων. Μας ενδιαφέρουν και θέματα επαναπρόθεσης. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω μία γενική εικόνα των εννέα χωρών που περιλαμβάνονται σε αυτό τον πυλώνα στον οποίο αναφέρομαι. Έχετε αυτό το γράφημα και να σας εξηγήσω, να σας πω τι κάναμε. Προσπαθήσαμε να κάνουμε απολογισμό, να δούμε τι έγινε και στις εννέα χώρες, στο σύνολό τους. Και αυτό απλά για να έχουμε έτσι μια ιδέα σε ποιον από τους τέσσερις πυλώνες έχουν εστιάσει τα προγράμματα και δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί. Πρέπει να σας πω, εκπλαγήκαμε από τα πορίσματα, γιατί είχαμε την εντύπωση ότι περίπου το 70% ασχολείται με την παράτυπη μετανάστευση και την ε, λαθροδιακίνηση. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Ε, το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε για περίπου το 30% που αντιστοιχεί σε αυτά τα δύο θέματα και στις εννέα χώρες. Στο δεύτερο πυλώνα αυτό έχει αρκετά ενδιαφέρον, αρκετό ενδιαφέρον. Μιλάμε για την υποστήριξη, μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση ε, και κινητικότητα και τα δύο ε, αντιστοιχούν στο 25% και ακολουθεί ο τρίτος ε, πυλώνας που είναι μεγιστοποίηση των προεκτάσεων της μετανάστευσης και της κινητικότητας στην ανάπτυξη. 11% είναι αυτό σε σχέση με την προστασία και τη χορήγηση ασύλου. Και εδώ επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε, άκουσα ότι αποδόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο καταπιστευματικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ότι ε, τα περισσότερα κονδύλια διατίθενται για τη διαχείριση των συνόρων. Αυτό λοιπόν το ταμείο και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το καταπιστευματικό ταμείο ε, αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε ανάλυση της κατανομής των κοντιλίων και διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό ε, των κοντιλίων από το Ταμείο που διοχετεύονται στην αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης, όχι απαραίτητα στη διαχείριση των συνόρων ή θέματα που έχουν καθαρά και μόνο σχέση με την ασφάλεια. μιλάμε για 42 εκατομμύρια που διατίθενται για τη διαχείριση των συνόρων. Όλα τα υπόλοιπα κονδύλια διοχετεύονται γενικότερα στην προστασία. Εδώ μπορείτε να δείτε ε, λεπτομερώς ε, τις ε, δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί. Δεν μιλάμε μόνο για χρήματα, μιλάμε και για πολιτικές δράσεις. Και βλέπετε εδώ την κατανομή στις ε, εννέα χώρες ε, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για Κινητικότητα. Βλέπετε εδώ διαφορετική κατανομή. Η Μολδαβία και το Μαρόκο έχουν αποφεληθεί περισσότερο από τις δράσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Μαρόκου ισχύει το εξής ότι υπάρχει μια ουσιαστική διμερή συνεργασία. Γι' αυτό βλέπετε αυτά τα αποτελέσματα. Τα κονδύλια που σχετίζονται με τη μετανάστευση, τα κονδύλια αυτά διοχετεύονται είτε μέσα από διμερείς συμφωνίες, είτε απευθείας από το κράτος μέλος. Αυτά τα οποία κάναμε ήταν να οργανώσουμε ε, τις κατηγορίες ε, με βάση κάποιες ε, λεπτομέρειες και προβήκαμε σε μία κοινή ανάλυση, ανάλυση την οποία κάναμε σε σχέση με τη Συμφωνία Κινητικότητας. Αυτά για όσους από εσά θέλετε να έχετε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχουν 50 πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί και αυτά απλά για να έχετε έτσι μια γενική εικόνα. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το εξής θελήσαμε να εστιάσουμε σε δράσεις που έχουν σχέση με τις επιστροφές. Και βλέπουμε εδώ ότι όσον αφορά τις 504 παρεμβάσεις στις 9 χώρες με τις οποίες υπογράψαμε συμφωνία, μόνο 17 δράσεις ε, σχετίζονται με επιστροφές. Διεπιστώνουμε λοιπόν Οι επιστροφές αυτές έλαβαν χώρα μόνο στις πέντε από τις εννέα χώρες. Έτσι, για να έχετε μια ιδέα περί τίνος πρόκειται. Τώρα, θα ήθελα με λίγα λόγια να εξηγήσω την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας κινητικότητας. Στην αρχή σας παρουσιάσαμε την ανάλυση που κάναμε και τώρα είμαστε σε μία ε, διαδικασία την οποία θα επεξεργαστούν περισσότεροι συνάδελφοί μας για να μπορέσουμε ε, τελικά να βελτιώσουμε το διάλογο με τις ε, χώρες που προανέφερα. Θα συναντηθούμε δηλαδή σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου και παράλληλα θα υπάρχουν και συζητήσεις τεχνικό επίπεδο για να περάσουμε στην πράξη. Τελευταία τώρα διαφάνεια. Όλα αυτά έχουν ως στόχο να συστήσουμε ένα είδος βαθμολογίου που θα αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συσταθεί ένας μηχανισμός ο οποίος θα επικαιροποιείται και αυτό ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε χώρας. Όσον αφορά τώρα τα ωφέλη, ε, θέλω να σας πω ότι προέκυψαν κάποια σημαντικά ωφέλη όπως ε, η υποστήριξη του νομοθετικού πλαισίου, αυξημένη κινητικότητα, ενίσχυση των δυνατοτήτων ε, των κρατών μελών και πρόοδος σε, θέματα θεωρήσεων. εμείς έχουμε ένα ιδιαίτερα πολύτιμο εταίρο και γι' αυτό έχουμε εδώ τους ε, συναδέλφους ε, οι οποίοι από τον οργανισμό ICMPD, τον κύριο Όλεκ Κυριτά, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας της ICMPD. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας αναπτύξουμε κάποια από τα συμπεράσματα σε ό,τι ε, αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών ε, κινητικότητας που υπό την αιγίδα της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής νέο, ε, νέα διευκόλυνση MPF Mobility Partnership Facility, όχι το ίδιο Migration Partnership Facility που, για το οποίο ακούσατε σήμερα το πρωί. Αυτό να το έχετε υπόψη σας καθώς θα ε, ε, μιλώ υπάρχει διαφορά. Είναι τα ίδια αρχικά αλλά άλλο πράγμα. Το πρόγραμμα αυτό της διευκόλυνσης χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και την ε, διευθύνουμε εμείς, ICMPD, για να κάνουμε τις συμφωνίες αυτές όλες όσο γίνεται πιο λειτουργικές. Βέβαια, πριν να μιλήσουμε για το ίδιο το πρόγραμμα, θα ήθελα να αναπτύξω λίγο κάποιες σημαντικές διαστάσεις του που συμβάλλουν στην εφαρμογή όλων των mobility partnerships και επίσης το πρόγραμμα MPF πώς στηρίζει τον υφιστάμενο τις υφιστάμενες δομές διαλόγου που έχουν δημιουργηθεί από τις Mobility Partnerships και το πρώτο έχει σχέση με, τα, με τους θεσμούς. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Mobility Partnership ως πλαίσιο συνεργασίας έχει περίπλοκο χαρακτήρα και ιδίω σε ό,τι αφορά το, τη διαδικασία διαλόγου που συνεπάγεται και βέβαια για την δημιουργία μορφών συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών μελών, οργανισμών και των χωρών που έχουν συνυπογράψει τις συμφωνίες αυτές. Για να στηριχτούν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι σημαντικό να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι φορείς από όλο το φάσμα για να σφυριλατηθεί μια πραγματικά ισχυρή εταιρική σχέση αλλά και πλέον αξιόπιστη. Σε ό,τι αφορά τις πρακτικές πτυχές οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας για παράδειγμα και οι νότιες χώρες. Βλέπουμε ότι στην Ανατολική Γειτονία το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο που συμβάλλει στην εφαρμογή των συμφωνιών είναι πιο στέρεο, πιο ισχυρό. Οι χώρες της Ανατολικής Γειτονίας έχουν κάνει προσπάθεια, για παράδειγμα, για να δημιουργήσουν δομές συντονισμού που θα επιτρέψουν την ορθή εφαρμογή των συμφωνιών και που δημιουργούν και παράγουν τα θετικά αποτελέσματα που επιθυμούν. Υπάρχουν, υπάρχει μια αρχιτεκτονική σε δύο βάσεις, αφενός τοπική πλατφόρμα συνεργασίας στην ίδια την χώρα, όπου ε, συμμετέχουν βεβαίως οι αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δεύτερο επίπεδο που έχει ο πολιτικό χαρακτήρα, δηλαδή με συναντήσεις υψηλού επίπεδου, που έχουν και μια πιο έντονη πολιτική διάσταση και συζητούν πώς θα προχωρήσει η Mobility Partnership. Ταυτόχρονα, όταν πρόκειται για τις δομές συντονισμού και τους θεσμούς, είναι σημαντικό να πει κανείς ότι, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, ότι όσο καλύτερος είναι ο συντονισμός για την εφαρμογή της Mobility Partnerships, τόσο καλύτερος είναι και, καλύτερη είναι και η ποιότητα του διαλόγου. Θα δείτε ότι μέσα στην Mobility Partnership Facility περιλαμβάνουμε τις σημαντικότερες και πολυπληθέστερες δράσεις στην Ανατολική Γειτονία. Αυτό πάλι απηχεί τον πιο ισχυρό στέρεο χαρακτήρα των θεσμών στις χώρες αυτές. Εξορισμού, mobility partnership σημαίνει ευθυγράμμιση και συντονισμό των διαφόρων προσδοκιών και συμφερόντων, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Η μετανάστευση, για παράδειγμα, είναι πάντοτε πολύ ευαίσθητο θέμα και περιλαμβάνει και πολύ ευαίσθητα θέματα όπως επιστροφές, όπως ε, προξενικές θεωρήσεις κλπ. Και όλα αυτά εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της MPF Partnership και πλήθος παραγόντων. Το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορούμε να κάνουμε να συνεργαστούν όλες, αυτοί, όλοι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι φορείς που είναι και φορείς διαφορετικών συμφερόντων. Πρώτα λοιπόν είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ε, μια κοινότητα στόχων και προσεγγίσεων σχετικά με την εφαρμογή της Mobility Partnership. Ταυτόχρονα να δημιουργηθούν κοινέ ευθύνε. Η Mobility Partnership θα πρέπει να βασίζεται σε διαφάνεια και σε υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη χρειάζεται από την αρχή, αλλά είναι και πολύ σημαντικό να δημιουργείται εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της συμφωνίας. Άλλο στοιχείο που πρέπει να σας απασχολήσει είναι πώς θα εξασφαλιστεί μια ισορροπημένη προσέγγιση για τη συνεργασία αυτή και να εξασφαλίσουμε και περισσότερη ισορροπία, για παράδειγμα, σε ξεχωριστές θεματικές περιοχές για την αντιμετώπιση των συμφερόντων των ε, χωρών εταίρων. Πρέπει να ε, εξεταστεί και η εξέλιξη των partnerships των ε, συνεργασιών αυτών, για παράδειγμα, για θέματα ασφάλειας. Όμως, εάν εξετάσει κανείς πάλι την, τις πρώτες mobility partnerships προδεκαετίας υπογράφηκαν αυτές, βλέπει κανείς ότι η στόχευση αλλάζει, διότι βεβαίως αλλάζουν και οι εθνικές προτεραιότητες και τα διάφορα ενδιαφέροντα των χωρών εταίρων. Αν μπορεί κανείς να εξετάσει από ψηλά όλες τις mobility partnerships, θα δει ότι περιλαμβάνουν θέματα μετανάστευσης, Ακούσαμε και τον εξοχότατο πρέσβη της Τινησίας που τόνισε τη σημαντική αυτή πτυχή. Είναι σημαντικό επίσης ότι από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και προστιθέμενες αξίες του πλαισίου Mobility Partnership συνολικά είναι ότι έχει συμβάλει στην δημιουργία συγκεκριμένων στρατηγικών για τη μετανάστευση από τις χώρες εταίρους. Και θα ήθελα να το τονίσω αυτό διότι χάρη στη σημαντική αυτή συμβολή τα ενδιαφέροντα και οι εθνικές προτεραιότητες των χωρών εταίρων ευθυγραμμίζονται πλέον με την ίδια την Mobility Partnership. Και από τότε που γράφηκαν οι συμφωνίες αυτές, Μολδαβία, Γεωργία, Πράσινο Ακροτήρι και άλλες χώρες έχουν εφαρμόσει τις πολιτικές αυτές. Η επόμενη διάσταση έχει σχέση με το γεγονός ότι η Mobility Partnership είναι εύκαμπτο όργανο και διεύκοντος μηχανισμό και αντιμετωπίζει όλα τα θέματα της μετανάστευσης με συνολικό τρόπο. Μπορεί λοιπόν να προσφέρει ένα πολύ ξεκάθαρο πλαίσιο και να επιτρέψει στους εταίρους να τοποθετούνται, να εκφράζουν ιδέες και προτεραιότητες, αλλά επίσης να θεσπίζουν συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή των ιδεών αυτών μέσω συγκεκριμένων έργων, project. Και τέλος, η τελευταία διάσταση αναφέρεται στο γεγονός ότι καταρχήν έχουν καινοτόμο χαρακτήρα οι mobility partnerships. Ορισμένες ε, χώρες εταίροι θεσπίζουν και καινοτόμα μέτρα, για παράδειγμα για την εμπλοκή της διασποράς, για την μετανάστευση και βεβαίως και ο ρόλος της Γενικής Διεύθυνσης ε, Home και του MPF είναι να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία, ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και ακόμα μεγαλύτερη κίνηση προς ακόμα περισσότερες mobility partnerships. Σε ό,τι αφορά το MPF ως πρόγραμμα και ως χρηματοδοτικό όργανο, ας το πω έτσι, μας ενδιαφέρει η κεφαλαιοποίηση των διδαγμάτων από την πράξη. Η Γκρατσιέλα προηγουμένως είπε ότι υπάρχουν άνω των 500 δράσεων που χρηματοδοτούνται και στηρίζονται από όλες τις Mobility Partnership και υπάρχει επομένως μεγάλος αριθμός συμπερασμάτων και διδαγμάτων που επιθυμούμε να κεφαλαιοποιήσουμε στο μέλλον. Χρειάζεται να ενοποιήσουμε βεβαίως έναν αριθμό σημαντικών στοιχείων των Mobility Partnerships και από την άποψη αυτή θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία συντονιστικών μηχανισμών από τις εννέα χώρες εταίρους μόνο δύο έχουν φτιάξει πλήρης μηχανισμούς συντονισμού όπως είπε και πριν η Γκρατσιέλα. Το MPF λοιπόν θα πρέπει να διαθέσει περισσότερες προσπάθειες προς το σκοπό αυτό. Να συνεχίσουμε εξάλλου να υποστηρίζουμε γενικά τη συνολική εφαρμογή και τον εννέα Mobility Partnership. Βλέπουμε βεβαίως ότι ορισμένες χώρες εταίροι εμπλέκονται περισσότερο, ισχυρότερα από άλλες θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στις προσπάθειες της ανατολικής και της νότιας γειτονίας. Να εξασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα επίσης και με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης διότι το MPF δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει μεγάλες δράσεις. Πρόκειται για στοχευμένες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις και από την άποψη αυτή χρειάζεται να συμβληθεί με άλλες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κατά βάση στο, το MPF χωρίζεται σε δύο σκέλη ας πούμε. Το ένα σκέλος προσφέρει επιχορηγήσεις σε χώρες μέλη για συγκεκριμένες δράσεις σε όλες και τις εννέα δηλαδή χώρες της mobility, των Mobility Partnerships. Υπάρχουν βέβαια τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες, αλλά θα τις αναπτύξω τώρα στα πλαίσια της παρούσας συζήτησης. Έχουμε ξεκινήσει μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τις χώρες μέλη μπορούν ανα πάσα στιγμή να καταθέσουν κάποια πρόταση, κάποιο σχέδιο που θα μπορεί να υλοποιηθεί σε μια συγκεκριμένη χώρα εταίρο Λίγα παραδείγματα ανατολικά, στην ανατολική γειτονία. Έξι δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται στην Αρμενία, η Γαλλία για παράδειγμα ε, κάνει εκεί ένα project για τις επιστροφές, η Σουηδία άλλο παρόμοιο σχέδιο, για παρόμοιο θέμα δηλαδή. Η Εστονία στην Γεωργία για διαδικασίες ασύλου. Η Ρουμανία έχει ολοκληρώσει μόλις ένα project για διαχείριση συνόρων με τη Μολδαβία. Και σε ό,τι αφορά τις νότιες χώρες, η Ιταλία έχει προχωρήσει ένα σχέδιο για την κυκλική μετανάστευση με την Ισία και Μαρόκο. Βλέπετε λοιπόν ότι το MPF είναι πολύ, ε, πολύ σχηδές σε ό,τι αφορά τα θέματα των οποίων επιλαμβάνεται. Επίσης και σε ό,τι αφορά τις χώρες εταίρους στις οποίες στοχεύουν οι δράσεις του. Τελευταία παρατήρηση είναι ότι έχουμε και ένα σκέλος το οποίο αναφέρεται στις διάφορες οριζόντιες διαστάσεις και μέσα στα πλαίσια αυτού έχουμε ξεκινήσει μια αξιολόγηση για τέσσερις mobility partnerships. Τα ξεκινήσαμε αυτά το 2008 και έγινε μόνο μια αξιολόγηση το 2012 για την εταιρική σχέση με την Μολδαβία. Γι' αυτό θεωρούμε σημαντικό τώρα να προχωρήσουμε την προσπάθεια αυτή για να δούμε ποια πράγματα έχουν επιτευχθεί μέσα σε μια δεκαετία περίπου mobility partnerships με συγκεκριμένες χώρες και να δούμε επίσης πώς λειτουργεί το πλαίσιο αυτό, η πλατφόρμα αυτής της συνεργασίας και πώς μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον. Όπως είπε η συνάδελφός μου Γρατσιέλα, του χρόνου θα οργανώσουμε μια εκδήλωση για να δούμε πώς εξελίχθηκε μέχρι τώρα ε, το MPF και πώς μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον. Έχοντας πει αυτά θα ήθελα ε, να σταματήσω εδώ και πολύ ευχαρίστω να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ και τον... Ε, θα δώσω μάλλον τώρα το λόγο και στους τρεις ε, ομιλητές, αφού προηγουμένως όμως ακούσουμε τις ερωτήσεις. Η κυρία Βερζιά. Κριστίν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους τρεις που πήραν το λόγο. Ε, στον κύριο Σερίφ θα αναφερθώ πρώτα δεδομένου ότι με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα του, η νησία. Θα ήταν καλό να ξέρουμε περισσότερα για το πώς έχει προχωρήσει η συμφωνία. Κατάλαβα που είπε ότι γίνονται συζητήσεις, αλλά δεν ε, έχω καταλάβει το εξή. Πρώτον, πιστεύω ότι μια πραγματική συνεργασία κινητικότητας πρέπει να βασίζεται και στην εταιρική σχέση και στην ισορροπία Άκουσα τις επιφυλάξεις σας και γνωρίζω ότι το θέμα έχει να κάνει κυρίως με την επιστροφή, την επανεισδοχή υπηκών τρίτων χωρών. Άκουσα επίσης ότι υπογραμμίζεται αυτό που θα έλεγα εγώ ελευθέρωση των θεωρήσεων για διαμονή μικρής διάρκειας. Πράγμα που δείχνει αυτό που όλοι ξέρουμε ότι αυτοί, αυτού του είδους οι θεωρήσεις δεν αλλάζουν τίποτα στην κατάσταση. Το είδαμε στα Βαλκάνια που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα από ότι οι χώρες Μαγκρέπ. Ετοιμάζουμε αυτή την εποχή το αίτιας. Όχι με τη δικιά μου σύμφωνη γνώμη, θα γίνει όμως παρόλα αυτά αυτό που ονομάζω εγώ χαμηλού κόστους θεωρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, με φύ τρόπο από την, την Ισία. Επίσης θα ήθελα να μας πείτε πιο συγκεκριμένα τι γίνεται με τους τινήσιους φοιτητέ. Με εκπλήσουν οι στατιστικές που διαβάζω για ολόκληρη την Αφρική και κυρίως αφορούν το Μαγκρέπ. Και φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι βορειοαφρικανοί φοιτητέ έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ξέρω, είμαι Γαλλίδα και βέβαια πρώτα απ' όλα τη Γαλλία επιλέγουν οι φοιτητέ αυτοί. Η κατάσταση δεν είναι ακόμα τραγική, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η γνώμη σα για αυτό το θέμα. Και εδώ για να επανέλθουμε και στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, ποια είναι η διεθνή εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Το ότι οι φοιτητέ αυτοί απεριμόνουν, ας πούμε, να μην πω απεριμόνουν, αλλά όλο και λιγότερο πάνε για σπουδές στις ε, χώρες ε, της Ευρώπης δεν είναι καλό. Λοιπόν, θα ήθελα περισσότερες ε, διευκρινήσεις. Και όταν ήμασταν στην Τινησία, συναντήσαμε υποσαχάριους μετανάστες στην Τινησία, και πολλοί από αυτούς μας εξήγησαν ότι δεν μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους διότι τους επιβάλλονται πρόστιμα, πολύ βαριά και αυτά είναι που τα εμποδίζουν να φύγουν. Οπότε εδώ δεν βλέπω συνοχή. Πώς γίνεται να εμποδίζεται με αυτόν τον τρόπο οι πικός τρίτων χωρών να επιστρέψουν στις χώρες τους. Και τώρα για συνολικά την μεταναστευτική αυτή συνεργασία. Εγώ δεν την καταλαβαίνω με την Λευκορωσία που είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει συμφωνία, κάνει, διαπραγματεύεται συμφωνία με τη χώρα αυτή. Εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι. Καταλαβαίνω ότι είναι αλακάρτ, ε, ελαστικές, προσαρμόσιμες και τα λοιπά τέτοιου είδου συμφωνίε που δεν έχουν καμία σχέση με συμφωνίε με άλλε χώρε, αλλά τι είναι αυτό το οποίο δικαιολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι Πολωνία, κάνει τέτοια συμφωνία κινητικότητας με τη Λευκορωσία. Για ποιες ροές μιλάμε εδώ και ποιες είναι οι ενδιαφερόμενες χώρες και τι κέρδος είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση μια τέτοια ε, συμφωνία. Και αυτό που ρωτάω ισχύει βέβαια και για όλες τις συμφωνίες. Γιατί αυτό στο οποίο έχω καταλήγω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά υποκαθιστά τις χώρες μέλη και στη θέση των χωρών μελών κάνει πράγματα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια προστιθέμενη αξία σε αυτό. Μα κανένα επιπλέον κέρδος. Και ζητάμε τελικά από το καταπίστευμα, το κατευθυντικό ταμείο, να υποκαθαστήσει την ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό λέμε. Δεν λέμε ότι ασχολείται κυρίως με την πολιτική ασφάλεια, λέμε ότι μέρος της πολιτικής ανάπτυξης μέσω του καταπιστωτικού ταμείου πηγαίνει για θέματα ασφάλειας. Είναι χρήματα δηλαδή που παίρνουμε από το αναπτυξιακό ταμείο, τα βάζουμε στο καταπιστωτικό ταμείο και τα χρήματα αυτά δεν πηγαίνουν για την ανάπτυξη. Σύμφωνοι, το ταμείο αυτό κάνει πολλά για την ανάπτυξη, αλλά χρησιμοποιούμε χρήματα μέσω αυτού του Αναπτυξιακού Ταμείου και δεν θα έπρεπε. Επίσης δεν κατάλαβα το Facility Program τι παραπάνω προσφέρει από το πρόγραμμα κινητικότητας. Σα είπατε ότι πρέπει να διακρίνουμε αυτά τα δύο και δεν κατάλαβα γιατί ίσως εγώ να μην ξέρω καλά το θέμα. Τέλος, Πρόεδρε, και θα τελειώσω με αυτό. Είδα όλους τους πίνακε στατιστικά, 105 δράσει κλπ. Πάρα πολύ ωραία. Καλό θα ήταν όμως να έχουμε μια πραγματική συνάντηση εργασίας για να δούμε αναθέμα όλες αυτές οι δράσεις τι σημαίνουν, γιατί ωραίοι πίνακες, αλλά ο καθένας ό,τι θέλει καταλαβαίνει. Τι σημαίνει αριθμός δράσης, εντάξει τι σημαίνει όμως για ποσά, στη χρηματοδότηση, τα κτλ. Ελπίζω να με στηρίξετε πρόεδρε. Δεν με ακούτε όμως. Πρόεδρε, φοράτε ακουστικά, μ' ακούτε. Α, τα έχετε τα ακουστικά, εντάξει. Εντάξει και... Τα γαλλικά μου έχουν βελτιωθεί τόσε φορέ που έχω πάει στη Γαλλία, λέει ο πρόεδρο. Ναι, ναι, όχι, είναι για να με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, έλεγα ότι πρέπει να κάνουμε μια πραγματική συνάντηση εργασία με του συναδέλφου που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Τέτοιο debriefing χρειάζεται για αυτού του πίνακε αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτό τι είναι μια πραγματική δουλειά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση και να ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδράση και αναχώρα. Ευχαριστώ. Μα κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει αυτά που λέτε κυρία Βερζιά. Βεβαίως και σας παρακολουθώ. Να δώσω το λόγο, κύριος Πολέζη. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, πρέσβη ο οποίος ε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε σε μια συμφωνία με την ε, Ιταλία για, τον, για την αγορά εξοπλισμού. Τι ήταν αυτό. Υπήρξε οικονομική συμμετοχή εκ μέρους της Ιταλίας. για Θα αρχίσω από τα πιο εύκολα, με το 2011 μετά τους 25.000 Ίσιους που πήγανε Λαμπαντούσα και μετά αλλού. Πρόκειται για 200 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία πήραμε εξοπλισμό για τα σύνορα, δηλαδή σκάφη, οχήματα κλπ. Πράγμα το οποίο μας βοήθησε να ανανεώσουμε τον ε, εξοπλισμό μας ε, για την προστασία και την ασφάλεια. Στη συνέχεια υπήρξαν εθελοντικά επιστροφές. Είχαμε συμφωνία για 30 περίπου άτομα κάθε εβδομάδα. Μετά θελήσαμε να αυξήσουμε τον αριθμό. Οι περισσότεροι από τους 25.000 επέστρεψαν λοιπόν στην Τινησία, οι περισσότεροι από αυτούς σε εθελοντική βάση. Δυστυχώς παραμένουν κάποιες εκατοντάδες σε κέντρα, σε καταβλισμούς και εδώ στο Βέλγιο για παράδειγμα. Καμιά εκατοστή. Ο υπουργό, πώς τον λένε. Α, ναι, ο κύριος Φράγκεν. Με ρώτησε, δεν μπορούμε να τους βάλουμε σε ένα αεροπλάνο όλους και να τους επιστρέψουμε. Και εγώ του είπα, όχι, δεν γίνεται. Γιατί πολλοί από αυτούς λένε ότι είναι την ίση χωρίς να είναι αν επιβεβαιωθεί από τα δαχτυλικά αποτυπώματα κτλ, τότε εντάξει. Αλλιώ, όχι. Ε, δεν είναι, να τους βάλουμε όλους μαζί και να μου φτιάξετε μια δεύτερη επανάσταση στην Τινησία. Όχι, να μου λείπει. Κύριε Βεζιά, τώρα όσον αφορά τους φοιτητέ, ξέρετε, υπάρχει μεγάλη δυσκολία για θεωρήσεις. Εξαρτάται και από τη χώρα. Και ίσως γι' αυτό μειώθηκε ο αριθμός των την θητητών στο εξωτερικό. Στη Γερμανία είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι στη Γαλλία. Αλλά υπάρχουν και πολλά πανεπιστήμια, ευρωπαϊκά, αμερικανικά και οι Ιαπωνέζικα μάλιστα για τους πιο λαμπρούς. Οπότε τι κάνουν, έρχονται στα πανεπιστήμια της Τινησίας και μας τους παίρνουν. Είναι κρίμα βέβαια για την Τινησία, γιατί εκεί οι δυνατότητε επιστροφή είναι δύσκολε. Αν κάποιο βρει μια καλή κατάσταση στην Ευρώπη ή αλλού, γιατί να γυρίσει στην Τινησία. Όσον αφορά του Αφρικανού μετανάστε, εγώ δεν έχω ιδέα για τα πρόστιμα αυτά που λέτε. Συγγνώμη που δεν μπορώ να σα απαντήσω, αλλά εγώ αυτό δεν το γνωρίζω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ήταν συναντήσεις που γίνανε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ακούσαμε τέτοια στοιχεία και τέτοια δεδομένα. Είχαμε μια τόσο καλή επίσκεψη στην Τινησία με την αποστολή μας. Πρέπει να σας ευχαριστήσουμε όλοι οι συνάδελφοι, γιατί εκεί μπορέσαμε σε βάθος να καταλάβουμε τι γίνεται. Καταλαβαίνουμε ότι η χώρα σας βρίσκεται υπό αλλά και ο κόσμος υποφέρει αναγνωρίζεται αυτό. Λοιπόν, τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε μπορούμε να σας τα παρουσιάσουμε όσον αφορά τα πρόστιμα. Όπως είπε και η κυρία Βερζιά και το ξέρει, κάποιοι βοηθούνται από οικογένειες στην Τινησία, αλλά περισσότεροι δυσκολεύονται με γραφειοκρατικές δυσκολίες κλπ. Θα σας τα δώσουμε τα στοιχεία. Ωραία. Ε, τώρα οι άλλοι η κυρία Ρίτσα πρώτα. Σύντομο όμως παρακαλώ, ε, δύο λόγια. Ναι, ευχαριστώ. Δύο πράγματα σύντομο. Όσον αφορά την εντολή για την ε, συνεργασία όσον αφορά την κινητικότητα, τα θέματα αυτά επικεντρώθηκαν περισσότερο σε ζητήματα ασφάλειας αλλά μπορώ για το συγκεκριμένο που με ρωτήσατε να ρωτήσω και εγώ τις υπηρεσίες μου και να σας στείλω την ε, αιτιολόγηση. Για το δεύτερο που ρωτάτε, για την στήριξη της διαχείρισης των συνόρων. Υπάρχουν αυστηρά κριτήρια από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς που ακολουθούν οι συνάδελφοι και αυτού του είδους η χρηματοδότηση εμπίπτει σε παλιότερο τίτλο. Άλλοι συνάδελφοι από τις άλλες υπηρεσίες ίσως είναι καλύτερα σε θέση να απαντήσουν. Για το τρίτο, για τους πίνακες και τα αποτελέσματα. Εμείς ότι χωρίς πρόβλημα να έχουμε μια τεχνική συνάντηση, να σας εξηγήσουμε τη λογική που ακολουθούν. Πάντως περισσότερο πρόκειται για αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί. Οι περισσότερες δράσεις δηλαδή που αναφέρουμε έχουν να κάνουν με τον κανονικό προγραμματισμό που περνάει από τη διαδικασία διαβούλευσης. Αλλά αν έχετε ιδέες, κάτι που να μπορεί να μας βοηθήσει περισσότερο στην ανάλυση και στην όλη αρχιτεκτονική του χειρήματο, ευχαρίστω είμαστε ανοιχτοί σε μια επικοδομητική συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ και στην ιστοσελίδα θα την βάλουμε την ε, παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε, πρέσβη Σερίφ, που μας βοηθήσατε τόσο πολύ. Είναι πολύ σημαντικό όσο μας είπατε και από ό,τι καταλάβαμε θα έχετε και άλλες επαφές. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας και για όλα μας είπατε. Σας ευχαριστώ και σας αγαπητοί συνάδελφοι από την DG Home. Και περνάμε στο επόμενο και τρίτο πάνελ για σήμερα το πρωί, οπότε παρακαλώ τους επόμενους ομιλητές να έρθουν εδώ στο βήμα. Και αρχίζουμε πρώτα με τον Dragos. Στη συνέχεια ο κύριος ε, Λεγκέρι και μετά ο κύριος Λιούις. Σήμερα το πρωί πρώτη παρουσίαση. Έχουμε πολλούς ομιλητές σήμερα το πρωί, είδατε. Και ευχαριστώ ήδη όλους όσοι συμμετείχαν. Τρίτο πάνελ λοιπόν, να σας παρουσιάσω τους επόμενους ομιλητές μας. Το θέμα μας είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα που είναι η πολιτική επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν διάφορες ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συστάσεις όσον αφορά μια πιο αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για επιστροφές. Η τελευταία της 27 Σεπτεμβρίου παρουσιάζει ένα χειρίδιο επιστροφών για τις χώρες μέλη και τις αρμόδιες αρχές τους προκειμένου να βοηθηθούν. Το Κοινοβούλιο πολλές φορές μέχρι σήμερα με ψηφίσματα του έχει ζητήσει την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τις επιστροφές. Ξέρετε ότι η θέση του Κοινοβουλίου είναι ότι η επιστροφή μπορεί να γίνει μόνο σύμφωνα με τους νόμους και τα δικαιώματα και μόνο σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς. Αυτά είναι τα κριτήρια για μας, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Γι' αυτό και θα θέλαμε να ακούσουμε τους ομιλητές μας και να έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στη συνέχεια για το θέμα. Ο πρώτος μας προσκεκλημένος είναι ο Τράγκος Τσουντοτσέ, λοιπόν, ο οποίος είναι τμήματάρχης για την παράτυπη μετανάσταση και την πολιτική επιστροφών. Καλώς ήρθατε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η πολιτική επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή η πολιτική καθορίζεται από πολλούς και περίπλοκους παράγοντες ε, ε, που έχουν σχέση και με τις τρίτες χώρες και με χώρες ε, διαμετακόμισης. Ε, σε αυτό το πάνελ αλλά και σε άλλες συζητήσεις ε, που έγινε συζήτηση για συνεργασία με άλλες χώρες νομίζω ότι συζητήθηκε σε βάθος πως το εξωτερικό κομμάτι η συνεργασία με τρίτες χώρες για τις επιστροφές πώς προχωράει όλη αυτή η κατάσταση την προηγούμενη εβδομάδα ε, σας έγινε ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, επιστροφές, τις μη δεσμευτικές συμφωνίες που έχουμε υπογράψει και γνωρίζω επίσης ότι υπάρχει και από αυτού μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Ε, και στην προηγούμενη εβδομάδα, αλλά ε, και με τον κύριο Αβραμόπουλο, έχουμε επισημάνει ότι τις επιστροφές τις θεωρούμε ως ένα κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτικής μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο ε, συνδέει την πράξη αυτή με επίδειξη αλληλεγγύης γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν μετανάστες που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να παραμείνουν στα κράτη-μέλη. Ε, βέβαια, εστιάζετε εσείς κυρίως ε, στο θέμα της εξωτερικής διάστασης των επιστροφών. Εγώ στη δική μου την ομιλία θα εστιάσω περισσότερο στην εσωτερική διάσταση, δηλαδή το τι ακριβώς σημαίνει στα κράτη-μέλη και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διάφορους οργανισμούς. Ας ξεκινήσουμε με το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ξέρετε ότι το 2008 εκπονήθηκε μία οδηγία που ορίζει τον κοινό παρονομαστή και τις διαδικασίες για να διασφαλίζονται οι κανόνες σε εθνικό επίπεδο για οτιδήποτε έχει σχέση από τον καθορισμό των συγκεκριμένων επιστροφών μέχρι και την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων. Εσείς στην Επιτροπή αυτή ξέρετε καλύτερα από τον καθένα ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν εύκολες, ότι χρειαστήκαμε πολύ χρόνο για να καταλήξουμε στο κείμενο της οδηγίας, αλλά από το 2008 έχουμε αυτή τη βάση για το πώς πρέπει να λειτουργούν επιστροφές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως θεματοφύλακας αυτού του πλαισίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλησε να ασχοληθεί με πρακτικές λύσεις, ε, με την υιοθέτηση της οδηγίας ε, από πλευράς κρατών μελών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Σέγγεν έχουμε κάνει και τις δικές μας αξιολογήσεις και καταλήξαμε στο εξής. Το 2015 κάναμε αξιολόγηση του Σέγγεν, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Λίχτενστάιν και για αυτές τις ε, συγκεκριμένες έρευνες ε, έχουν υποβληθεί και προγράμματα δράσεις έχουμε ήδη καταλήξει ε, στην τελική μας αξιολόγηση. Το 2016 είχαμε αποστολές στο Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Μάλτα και Γαλλία και άλλες δύο έχουν ανακοινωθεί ε, στο Καλέ, στη Γαλλία, όπως επίσης και στη Γερμανία. Σε όλες λοιπόν αυτές τις ε, αποστολές, εκτός από αυτή της ε, Γερμανίας, ε, ήδη είμαστε στη φάση της εφαρμογής συγκεκριμένων προγραμμάτων και εμείς προβαίνουμε στη δική μας την αξιολόγηση. Το 2017 είχαμε αποστολές στη Δανία, Ισλανδία, Σουηδία, Πορτογαλία, Ισπανία και Νορβηγία για αξιολόγηση του Σέγκεν και άλλη μία χωρίς ανακοίνωση στην Ουγγαρία για να δούμε τις συνθήκες κράτησης οι αξιολογήσεις και οι εκθέσεις αυτών των αποστολών του 2017, αυτές ακόμα βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας. Για το 2018 θα επισκεφτούμε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, ε, την Σουηδία, Λετωνία, Λιθουανία, Φινλανδία και έτσι θα ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο αξιολόγησης ε, των κρατών που συμμετέχουν στη Συμφωνία Σέγγεν. Σε τρία χρόνια θέλουμε να έχουμε επισκεφτεί όλα όλα τα κράτη να έχουμε μία βάση για να μπορούμε να αξιολογήσουμε πώς ακριβώς εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές σε εθνικό επίπεδο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια ε, λαμβάνουν τις εκθέσεις μας και για τις προγραμματισμένες και για τις ε, ξαφνικές επισκέψεις. Ε, το Δεκέμβρη ε, στην Επιτροπή, Υποεπιτροπή του Σέγγεν και κλεισμένων των θυρών μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το περιεχόμενο της δουλειάς μας κατά διάρκεια αυτών των επισκέψεών μας. Αυτό θα το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η σύσταση που ενέκρινε η Κομισιόν το Μάρτιο του 2017, ο πρόεδρος το είπε ήδη, κατά την άποψή μας είναι ένα σημαντικό έγγραφο, διότι και εμείς, όπως σας είπα, μπορέσαμε να βασιστούμε στις αξιολογήσεις επισκέψεων σε χώρες Σέγγεν, να εστιάσουμε σε πορίσματα και να υποβάλουμε προτάσεις στα κράτη-μέλη για το πώς μπορούν τα μέτρα και την ομοθεσία τους να τα προσαρμόσουν καλύτερα στην διοικητική πρακτική. Βασικός μας ε, στόχος είναι να επιτύχουμε μεγαλύτερη διοικητική συνοχή με βάση αυτά που ανακαλύπτουμε στα κράτη-μέλη. Γιατί βλέπουμε ότι τα προβλήματα προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση. Επίσης, ε, στη διάρκεια ή κατά τη διάρκεια εκπόνηση συστάσεων ε, θελήσαμε να ασχοληθούμε με τις ε, συνθήκες κράτησης επίσης και με την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των κρατουμένων με βάση τις υπάρχουσες συμφωνίες. Θέλουμε μια πιο ενιαία ρύθμιση για υποβοηθούμενες επιστροφές Επίσης επιθυμούμε να επιτύχουμε καλύτερη χρήση ε, όλων αυτών που προβλέπονται στην οδηγία. Ε, τα κράτη-μέλη έλαβαν υπόψη τους ε, τη σύσταση και προέκυψε ε, ένα πρόγραμμα για το πώς ακριβώς τα κράτη προτίθενται να εντάξουν τις συστάσεις στην πρακτική τους. Ανακοινώθηκε άλλο ένα βήμα, δηλαδή με την ε, έγκριση και υιοθέτηση του εγχειριδίου για τις επιστροφές. Αυτό ήταν ένα κομμάτι της ανακοίνωσης του 2017. Νομίζω όλοι γνωρίζετε ότι ορισμένα κράτη-μέλη είπαν από τις αρχές του έτους και ορισμένα μάλιστα και αργότερα ότι ότι επιθυμούν τροποποίηση της οδηγίας για τις επιστροφές. Εμείς ως Κομισιόν είμαστε κατά της ε, τροποποίησης αυτής της οδηγίας γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι μπορεί να επιτευχθεί με τους ισχύρτες κανόνες ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών στο βαθμό που τα κράτη-μέλη είναι πρόθυμα να κάνουν καλύτερη επένδυση ε, και καλύτερη, καλύτερο συντονισμό. Ε, είδαμε πώς λειτουργούν τα περισσότερα συστήματα, τα εθνικά συστήματα και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν εμπέλτες πρακτικές στα κράτη-μέλη που δείχνουν ότι ό,τι συστήνουμε στις Βρυξέλλες ε, ε, μπορεί πράγματι να εφαρμοστεί. Απαιτούν όλα αυτά προσπάθειες, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχει η βάση. Ας πάμε τώρα στο ε, εφαρμοστικό εργαλείο ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ανακοίνωση της 27 η Σεπτεμβρίου εντοπίζει και άλλο ένα σημαντικό παράγοντα για τις επιστροφές. Πρόκειται για τον Ευρωπαϊκό Φορέα Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Είμαι σίγουρος ότι ο συνάδελφός μας θα σας ενημερώσει επ' αυτού. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε αποδώσει σημασία στο ρόλο αυτής της υπηρεσίας ε, διότι έχουμε καταλήξει στο ότι ο ρόλος αυτός είναι σημαντικός. Πρέπει να πούμε ότι ο φορέας της συνοριοφυλακής και της ακτοφυλακής έχει συμβάλει πάρα πολύ. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία που το τεκμηριώνουν. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, διότι είμαι σίγουρος ότι ο ε, διευθυντής ε, της υπηρεσίας θα σε ενημερώσει καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά στο μέλλον. Ε, στο μέλλον, λοιπόν, και σε σχέση με την πολιτική των επιστροφών, αυτή ε, σχετίζεται με την ευρύτερη πολιτική μετανάστευσης. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Ό,τι κάνουμε για τα θέματα αλληλεγγύης και ασύλου επηρεάζουν και το πώς τροποποιούμε, αν κριθεί απαραίτητο, την πολιτική μας των επιστροφών. Οι επιστροφές θα συνεχιστούν, όπως ήδη συζητήθηκε σήμερα το πρωί, θα συνεχίσουν να είναι άμεσα συνδεμένες με την εξωτερική πολιτική, με τη συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διαμετακόμισης. Ε, θα ενημερωθείτε για τις εξελίξεις με την τελευταία έκθεση που εγκρίναμε πριν από δύο εβδομάδες. Έχουμε σταθεροποιήσει ε, τα διάφορα στοιχεία της μετανάστευσης γιατί θέλουμε θέλουμε να μπορούμε σε τακτική βάση να ενημερώνουμε, να έχουμε μια ε, γενικότερη άποψη των δράσεων που υλοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Okay, we'll take those questions at the end of the panel. Um, next we have um, Fabrice Legeri, who we all know, of course, Executive Director of the European Border. Ο επόμενος ομιλητής, παρακαλώ, που είναι εκτελεστικός διευθυντής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ βεβαίως και τις αξιότιμες και αξιότιμους κύριους Ευρωβουλευτές για την ευκαιρία που μου δίνετε να αναπτύξω για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή. Όπως τονίστηκε από τον κύριο Τιντοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πολιτική επιστροφών είναι μία συνιστόσα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή έχει νέες αρμοδιότητες από πέρσι. Μπορώ να σας δώσω ορισμένα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Ο αριθμός πτήσεων επιστροφών που οργάνωσε ο οργανισμός μας φέτος έχει ξεπεράσει τις 300 ο αριθμός παράτυπων μεταναστών που επεστράφησαν με την υποστήριξη του οργανισμού μας έχει φτάσει ήδη 2.500, στις 2.500 φέτος πέρσι ολόκληρο το χρόνο ο οργανισμός υποστήριξε τις χώρες μέλη για τις επιστροφές 10.700 παράτυπων μεταναστών και 232 πτήσεις. Αν συγκρίνουμε τους αριθμούς αυτούς με αυτούς του 2015, είναι ακόμη πιο προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τι αυτή έχει αναπτύξει πολιτική επιστροφών και έχουμε πολλαπλασιάσει, έχουμε πενταπλασιάσει το λιγότερο τα υλοποιήσιμα από πλευράς οργανισμού. Όμως θα πρέπει να επαναλάβω και πάλι ότι η απόφαση για επιστροφή, η απόφαση περί επιστροφής είναι εθνική υπόθεση. Μόνο οι εθνικές αρχές, μόνο οι χώρες μέλη μπορούν να αποφασίσουν ποιος θα επιστραφεί. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Υπάρχει ανάγκη μιας ενίας ευρωπαϊκής πολιτικής, όπου οι χώρες μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και η Ακτοφυλακή θα συνεργάζονται στενά. Έχουμε σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές δραστηριότητες υποστήριξη ταυτοποίησης θα επανέλθω μετά σε αυτό γιατί μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η ορθή ταυτοποίηση του μετανάστη για να μπορέσουμε να καθορίσουμε ποια είναι η χώρα προέλευσης και για να λάβουμε τα ταξιδιωτικά έγγραφα από την χώρα προορισμού. Από τη χώρα μάλλον προέλευσης, διορθώνω. Ο οργανισμός μας προβλέπει μετακίνηση με αεροσκάφη που διαθέτουν οι χώρες μέλη, αλλά τώρα Βρισκόμαστε σε διαδικασία υποβολής προσφορών και σύντομα από τον Ιανουάριο ο οργανισμός μας θα μπορεί να αναβλώνει αεροσκάφη από μόνος του. Στα πλαίσια της ε, δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας υποστηρίζει ο οργανισμός και μενάβλωση οχηματαγωγών για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών μέχρι τώρα το 2017 μεταφέρθηκαν 650 πρόσωπα από τα ελληνικά νησιά προς την Τουρκία από την Frontex στα πλαίσια της δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Επίσης, και αυτό είναι σημαντικό, διεξάγονται στρατηγικής φύσης συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προτείναμε στι χώρες μέλη κάποιε επιχειρησιακές δράσεις ώστε να ενισχύσουμε την συνεργασία, την τριγωνική αυτή συνεργασία χώρες μέλη, κομισιόν και οργανισμός μας. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία της τριγωνικής αυτή σχέσης είναι η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Εθνικών Αρχών Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οργανισμού μας που θα πρέπει να ενισχυθεί. Εάν, για παράδειγμα, ο οργανισμός συνοφυλακή ακτοφυλακής μπορεί να οργανώσει και να σχεδιάσει από μόνος του πτήσεις τσάρτερ θα πρέπει ο οργανισμός να γνωρίζει ποιοι είναι οι προορισμοί και ποιος είναι ο σχεδιασμός. πότε θα πρέπει οι, οι, οι μετανάστες, πότε θα είναι έτοιμοι να επιστραφούν. Δεν λαμβάνει ο οργανισμός τις αποφάσεις αυτές, αλλά οι χώρες μέλη οφείλουν να κοινοποιούν τον αριθμό των προσώπων της εθνικότητας και ούτω καθεξής και της χώρες προορισμού βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα σύστημα πληροφορικής που λέγεται Ήρμα, να το θέσει δηλαδή στη διάθεση του οργανισμού φυλακή Ακτοφυλακή, Θα το επεξεργαστούμε αυτό και αυτό είναι και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του σχεδίου δράσεω που προτείνει ο οργανισμός. Διεξάγεται και μια συζήτηση στρατηγικής, έγινε μάλλον εχθές στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΑΣΟ γιατί μια άλλη πρόκληση στη διαχείριση του μεταναστευτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι ο αριθμός μεταναστών που υποβάλλουν αιτήσεις ασύλου είναι πολύ υψηλός. Ενώ ο αριθμός των προσώπων που τους χορηγείται τελικώς το άσυλο είναι πολύ χαμηλότερος. Οι άνθρωποι που δεν λαμβάνουν τελικώς το καθεστώς του ασύλου δεν λαμβάνουν και άδεια παραμονής. Και αυτό είναι ακριβώς το πεδίο εφαρμογής της επιστροφής. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση στρατηγικού χαρακτήρα με τον ΕΑΣΟ και με τις αρμόδιες εθνικές αρχές, αρμόδιες για το άσυλο, ώστε να είμαστε σε θέση να ανταλλάσσουμε καλύτερα πληροφορίες για τις απορριπτόμενες αιτήσει ασύλου, ώστε τα πρόσωπα των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε να μπορούν να εντάσσονται στο σύστημα επιστροφών. Εδώ βρισκόμαστε ως state of play. Να έρθω τώρα σε ένα άλλο θέμα που ίσως ενδιαφέρει περισσότερο στα πλαίσια της σημερινής ακροάσεως και που έχει σχέση με τη συνεργασία με τρίτες χώρες και πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις στο πεδίο των επιστροφών. Ο οργανισμός δρά υπό την αιγίδα της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής και αναφέρομαι στη στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων σε ό,τι, αφορά την εφαρμογή των συμφωνιών επιστροφών και συνήθως ο οργανισμός μας υποστηρίζει με εμπειρογνώμονες το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν αυτή διαπραγματεύεται συμφωνίες επανεισδοχής. Συμμετέχουμε επίσης και σε τακτικές συναντήσεις κοινών επιτροπών με τις ε, τρίτες χώρες. Έχουμε και συμφωνίες συνεργασίας που υπογράφει ο οργανισμός. Σε ορισμένες από αυτές περιλαμβάνεται και παράρτημα σχετικό με τις επιστροφές. Βλέπε συμφωνία με την Ιγυρία. Δεν είναι σύνηθες αυτό. Με την Ιγυρία όμως ο οργανισμός μπόρεσε προετών να αναπτύξει μια καλά ε, θεμελιωμένη συνεργασία. Συνεργαζόμαστε και με τον αξιωματούχο σύνδεσμο για τις επιστροφές των χώρων μελών, τους συνδέσμους δηλαδή. Έχουμε και αξιωματούχους συνδέσμους που θα μπορέσουν στο μέλλον να παίξουν ένα ρόλο στο πλαίσιο των επιστροφών. Επίσης, επιστροφές που οργανώνονται από τον οργανισμό εκτελούνται από τον οργανισμό αλλά οργανώνονται από τις χώρες προέλευσης, ιδίως τα Βαλκάνια. Και αυτό σημαίνει, είναι, εντάσσεται μάλλον στα πλαίσια μιας πολιτικής ανάπτυξης ικανοτήτων, capacity building, δηλαδή να μάθουν οι χώρες αυτές πώς να οργανώνουν τις επιστροφές, επιχειρήσεις επιστροφών, διότι και αυτές αντιμετωπίζουν προκλήσεις και αυτές οι χώρες οφείλουν να οργανώνουν πτήσεις επιστροφών, ιδίως όπως είπα χώρες των Βαλκανίων. Έχουμε και μια αποστολή ταυτοποίηση. δηλαδή ε, συνεργαζόμαστε με τις προξενικές αρχές για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων. Έχουμε κάνει τέτοιε identification missions στην Ιταλία. Έχουμε και βραχυπρόθεσμες σχετικές αποστολές σε διάφορες άλλες χώρες μέλη. Και θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι όλες αυτές οι δράσεις εκτελούνται σε απόλυτη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ιδίως δε ο οργανισμός έχει μια ομάδα αξιωματούχων που παρακολουθούν, monitor δηλαδή, ιδίως για τις επιστροφές μέσω πτήσεων και όλες τις συλλεκτικές πτήσεις. Από τη σκοπιά του οργανισμού είναι αναγκαίο να υπάρξει μια συνολική, μια ε, σε βάθος προσέγγιση, ένα ενοποιημένο σύστημα επιστροφών που σημαίνει ότι οι Εθνικές Αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για κάθε πτυχή της πολιτικής επιστροφών. Ο οργανισμός βεβαίως ενδιαφέρεται να έχει στη διάθεσή του επιχειρησιακά δεδομένα, αλλά χρειαζόμαστε επίσης μια ευρύτερη προσέγγιση όπως συζητήθηκε στην ακρόαση σας σήμερα το πρωί σχετικά δηλαδή με την ανάπτυξη η πτυχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ώστε να μην περιοριστεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών μονάχα σε μια πολιτική επιστροφών. Έχω υπόψη την μελλοντική νότια γειτονία που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε επίσης τα πλαίσια της ε, κοινότητας συλλογής πληροφοριών Frontex για συνεργασία με Αφρική. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ικανοτήτων των αφρικανικών χωρών να συνεργαστούν δηλαδή σε θέματα διαχειρίσεως των συνόρων που έχουν σχέση και με την ε, ασφάλεια στην Αφρικανική Ήπειρο. Αν θέλουμε λοιπόν μια αμοιβαία υποφελή προσέγγιση και, συμφωνώ, και ομιλώ βεβαίω εδώ για δραστηριότητες, για επιχειρησιακές δραστηριότητες πάντα μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του οργανισμού θα πρέπει να διευρύνουμε τα πεδία εφαρμογή και να περιλάβουμε και ζητήματα ασφαλείας τα οποία δεν άπτονται άμεσα της μετανάστευσης αλλά ωστόσο προκαλούν ανησυχία. Χώρες Σαχέλ για παράδειγμα που για αυτές η ασφάλεια είναι υπαριθμόν ένα ανησυχία. Χάρη στην ευρύτερη εντολή χάρη σε ε, συνεργασίες όπως η ΑΦΙΚ, African Intelligence Community, θα μπορέσουμε νομίζω να αναπτύξουμε τον διάλογο στα πλαίσια της διαχείρισης των συνόρων και με τις χώρες αυτές. Βεβαίως και υπάρχει ανάγκη μακροπρόθεσμης πολιτικής ανάπτυξης απέναντι στις χώρες αυτές. Όμως αυτό δεν εντάσσεται στο πεδίο δραστηριότητα του οργανισμού μας. Πάντως, από τη δική μου σκοπιά αυτό είναι απολύτω αναγκαίο. Δεν μπορούμε καν να εκτελέσουμε μια ορθή πολιτική επιστροφών αν δεν εξισορροπείται αυτή από μια πολιτική ανάπτυξη και ιδίω απέναντι στην Αφρικανική Ήπειρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τελευταίο ομιλητή του παρόντο πάνελ είναι ο κ. Μπεν Λιούι από το γραφείο του ΥΠΑ του Αρμοστού για του πρόσφυγε των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε. Θα είναι κάπως διαφορετική η δικιά μου παρουσίαση και η δικιά μου παρέμβαση. Δεν είμαι εμπειρογνώμων για ευρωπαϊκά ζητήματα, αλλά θα σας εκφράσω τις ανησυχίες του είπα του αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά τις μετακινήσεις μεταναστών, τις επιστροφές κτλ και όσον αφορά και τα νέα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιστροφές αυτές. Συχνά λέμε ότι οι επιστροφές είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει καλά ένα σύστημα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών. Πόσο θετικά ακούγεται αυτό για τόσο πολλές επιστροφές που ξέρουμε ότι τελικά δεν ανταποκρίνονται σε αυτή την όμορφη εικόνα. Αν κάποιος πρέπει να επιστρέψει, είτε το κάνει σε θελοντική βάση είτε καταναγκαστικά, πρέπει να ξέρουμε ότι πρόκειται για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να φεύγουν από μια επικράτεια. Και κάτι δεν έχει πάει καλά για να συμβαίνει αυτό, είτε όσον αφορά τα, τις ασφαλές μεθόδους μετανάστευσης ή γιατί δεν τα καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να ζήσουν στην καινούρια χώρα και αναγκάζονται να επιστρέψουν στην χώρα προέλευσής τους. Θέλω να είμαι και σαφής ευθύ εξ αρχής για το τι μιλάμε όταν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο επιστροφές. Ακούγεται έτσι κάπως γυμνός, αλλά πρέπει να τον βάζουμε στο συγκεκριμένο του πλαίσιο. Εμείς έχουμε ελέγξει κάπως τις πολιτικές επιστροφών και τις πρακτικές μάλλον αυτές και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτές τις πρακτικές και του χρόνου και εμείς καταλαβαίνουμε ότι είτε γίνεται η επιστροφή αυτή σε εθελοντική βάση είτε όχι πρόκειται για μια βία διαδικασία τουλάχιστον έτσι την εισπράττει ο ενδιαφερόμενος. Οι άνθρωποι αυτοί σπάνια επιστρέφουν με αξιοπρέπεια σε μια χώρα όπου γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματά τους η οποία αυτή η χώρα μπορεί να μην είναι καν δικιά του μερικέ φορέ. Οπότε η επιστροφή δεν είναι μια πραγματική επιστροφή, δεν επιστρέφουν από κάπου που φύγαν, πάνε σε μια άλλη χώρα που δεν είναι η δικιά του. Και πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί για την πραγματικότητα των ε, επιστροφών. Αυτέ οι επιστροφέ, ο όρο αυτό είναι μάλλον εφημισμό που περιγράφει κάτι διαφορετικό, που περιγράφει την επιστροφή ανθρώπων σε χώρες για λόγους ε, που ιστορικά τους έχουν εμποδίσει να έχουν πρόσβαση εκεί κανονικά. Οπότε, έχοντας αυτό υπόψη, ας μιλήσουμε τώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις επιπτώσεις τους. Πρώτον, ε, δεν επιτρέπεται ε, βία να μεταφέρει έναν άνθρωπο κάπου αλλού. Αυτό δεν είναι δικαίωμα. Και πάντα οποιαδήποτε δράση πρέπει να περιορίζεται από τόσα ισχύουν στις διεθνείς συνθήκες. Η, η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λέει ότι όλοι είναι ίσοι όσον αφορά την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, που σημαίνει ότι αν είναι να περάσουν κάποια σύνορα, η χώρα στην οποία βρίσκονται έχει υποχρεώσεις απέναντί τους, απέναντι σε όλους τους μετανάστες. Είτε έχουν ε, κάνει αίτηση για άσυλο, είτε έχουν άσυλο. Το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπει προστασία για όλους τους μετανάστες. Και όταν μιλάμε για δικαιώματα, εδώ υπάρχει κάποια αλληλεξάρτηση μεταξύ τους και είναι αδιέρετα. Δεν είναι επίσης αμοιβαία αποκλειόμενα. Που σημαίνει ότι πρέπει να χαίρουν των δικαιωμάτων που τους προσφέρουν οι διεθνείς συμφωνίες αλλά και οι ειδικέ συμφωνίες. Και αυτό ισχύει κυρίως στην Ευρώπη όπου από τη μια υπάρχουν οι πρόσφυγες οι οποίοι δικαιούνται διεθνή προστασία και όλοι οι άλλοι που θεωρείται στην Ευρώπη ότι δεν ε, πρέπει να χαίρουν τέτοιε διεθνούς προστασίε. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Όλοι υπόκεινται σε αυτό το δικαίωμα. Είτε πρόκειται για πρόσφυγε είτε και μετανάστες. Οι πρόσφυγες έχουν επιπλέον. Ή τα παιδιά έχουν επιπλέον δικαιώματα. Οι γυναίκε που έχουν δικαιώματα σε διαφορετικά πλαίσια. Οι εργασιακά δικαιώματα υπάρχουν. Οπότε είναι πολύ πιο περίπλοκο το ζήτημα από ότι να βάζουμε του πρόσφυγες από τη μια μεριά, τους σε άσυλο από τη μια μεριά και όλου του υπόλοιπου από την άλλη. Γι' αυτό και μιλάμε για τις διάφορες διαδικασίες, την εγγύηση δικαιωμάτων, τις ε, μετακινήσεις, τις ε, καταναγκαστικές επιστροφές κτλ. Είπα πριν ότι είναι αλληλένδετα τα δικαιώματα αυτά και αδιέρετα και ότι ο καθένας δικαιούται τις υψηλότερες προδιαγραφές δικαιωμάτων βάσει των διεθνών ε, συμφωνιών. Υπάρχουν νέα βασικά μέσα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι τουλάχιστον πρέπει να υποφελούνται από θεμελιώδη δικαιώματα, είτε πρόκειται ε, των πολιτών, είτε πρόκειται για οικονομικά, είτε για πολιτικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά. Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις, ούτε σε βάρος των γυναικών κλπ. Και υπάρχει και σύμβαση για τα εργασιακά δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικυρώσει και, τις, ε, και τα εννέα αυτά βασικά εργαλεία μέσα, οπότε είναι υποχρεωμένη και να τα σέβεται. Και συμβαλόμενες ε, σε τέτοιες διεθνείς συνθήκες, οι χώρες μέλη αναλαμβάνουν να σέβονται, να προστατεύουν και να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτές για όλους όσους βρίσκονται στην επικράτειά τους και να ελέγχουν ότι όντως γίνεται αυτό που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει ούτε να παρεμβαίνουν ούτε να περιορίζουν την απόλαυση τέτοιων ε, δικαιωμάτων μέσω των εξωτερικών τους ε, δράσεων ή πολιτικών. Αν εξετάσουμε τώρα τις ανησυχίες όσον αφορά τις πολιτικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστροφή. Τον, ε, στις 3 ε, Μαρτίου φέτος η υπηρεσία μας προέβησε κοινή δήλωση με τη UNICEF με την οποία εκφράζει τις ανησυχίες όσον αφορά τις νέες προτάσεις για πολιτικές επιστροφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέγοντας ότι πρόκειται για παραβίαση τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών για την μετανάστευση ότι δεν υπάρχει επαρκής προστασία των παιδιών και θα σας εξηγήσω και αργότερα και αν ενδιαφέρεστε περισσότερο υπάρχει συζήτηση μεταξύ της Επιτροπής Μεταναστών και Προστασίας των Παιδιών όπου εκεί αναφέρεται ότι η προστασία των παιδιών πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα πάνω από την μετανάστευση, τον έλεγχο των συνόρου και οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Στις 9 Μαρτίου επίσης μια ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών έκανε κοινή δήλωση για τις πολιτικές αυτές επιστροφών λέγοντας εδώ πέρα ότι πρόκειται για ολίσθημα και σημειώνει ότι αυτές οι προτάσεις μειώνουν τις δικλίδες ασφαλείας και ενθαρρύνουν ε, παραβιάσεις μέσω της ε, κράτησης των παιδιών και των οικογένειών τους ή ε, παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην ακρόαση που είχε γίνει εδώ πέρα τον Απρίλιο, πολλοί εδώ μέσα είχαν πει ότι οι συμφωνίες αυτές που γίνονται οδηγούν σε μια τάση την Ευρωπαϊκή Ένωση για περισσότερη πίωση και ε, καταναγκαστικές ε, επιστροφές που απομακρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα περισσότερο από τις ίδιες τις αρχές της. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν τα κενά αυτά που έχουμε διαπιστώσει στα πλαίσια της μεταναστευτικής ε, διαχείρισης, η υπηρεσία μας δημοσίευσε το 2014 συστάσεις για κατευθυντήριες ε, γραμμές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα διεθνή σύνορα. Βασιζόμαστε στα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το πώς να τηρήσουμε περισσότερο τις υποχρέσεις μας απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Υπάρχουν 10 κατευθυντήριε γραμμέ, πολύ συγκεκριμένε, που βοηθούν τι χώρε μέλη να παίρνουν μέτρα προστατεύοντα τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο τέτοιε κατευθυντήριε γραμμέ. Πρόκειται για τις ε, επιστροφές που δεν πρέπει να είναι βίες. Πρώτα απ' όλα, η κατευθυντήρια γραμμή είναι, λέει ακριβώς αυτό, ότι οι επιστροφές, η μετακίνηση των μεταναστών δεν θα πρέπει να γίνεται βία, ε, θα πρέπει να τηρείται η αρχή της μη επαναπρόθεσης του νορεφουλμό και να μην γίνονται αυθαίρετα συλλογικές ε, απελάσεις. Δεν έχω βέβαια καιρό να μπω σε όλες τις λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία μόνο θα σας δώσω. Όσον αφορά ακριβώς την αρχή του νορεφουλμό, της μη επαναπρόθεσης. Αυτό είναι κάτι επιτακτικό, μια επιτακτική ε, προδιαγραφή του διεθνούς δικαίου που επεκτείνεται πέρα από τους μετανάστες ή τους πρόσφυγες. Είναι κάτι που ισχύει ως διεθνές δίκαιο μαζί με την απαγόρευση βασανισμών, κακομεταχείρισης ή άλλοι ανήκε στο βλάβη. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος υποβάλλεται σε επιστροφή δεν πρέπει να υποφέρει από τέτοιου είδους ε, κακοποίησης Είτε καλύπτεται το καθεστώς ασύλου, είτε όχι. Επίσης υπάρχει το θέμα της δέουσας νομικής διαδικασίας, η οποία πρέπει να τηρείται και οι μετανάστες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν ένδικα μέσα εφόσον το επιθυμούν να έχουν και την ευκαιρία να το κάνουν εφόσον θέλουν. Και επίσης δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, να τους εξηγούμε γιατί έχει ληφθεί η απόφαση αυτή για να επιστρεφούν, σε γλώσσα που να καταλαβαίνει ο ενδιαφερόμενος και που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει δωρεάν διερμηνία κλπ. Τέλος, οι διαδικασίες επιστροφής θα πρέπει να ελέγχονται από έναν εξάρτητο σώμα, δηλαδή να υπάρχουν αρχές οι οποίε να είναι ανεξάρτητες από τις αρχέ οι οποίε προβαίνουν στι επιστροφέ αυτές και να μπορούν να επιβλέψουν την όλη διαδικασία για να δουν κατά πόσο τηρούνται οι κανονισμοί. Περνάω τώρα στην κατευθυντήρια γραμμή αριθμό 10 για τη συμφωνία συνεργασία. Εδώ ξέρουμε ότι κάθε διασυνοριακή συνεργασία πρέπει να βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, να δίνει εγγύσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό εμείς προτείνουμε αυτή την προσέγγιση βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σημαίνει ότι οι συμφωνίε δεν θα πρέπει να γίνονται με χώρε οι οποίες δεν μπορούν να αποδείξουν ότι μπορούν να προστατεύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η προσέγγιση βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να έχει να κάνει με διάφορα δικαιώματα και να συμβάλλουν σε αυτό όλε οι αρχέ και αυτέ οι μόρφωσες του νόμου και όχι. Όσες ε, δεν έχουν τέτοια εντολή σεβασμό τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούν ε, να συμπεριλαμβάνονται. Πρέπει επίσης ε, να αξιολογούμε τα αποτελέσματα, κατά πόσο τηρούνται οι προδιαγραφές. Οι συμφωνίες συνεργασίας αυτές καθεαυτές πρέπει να ελέγχονται λοιπόν και να υπάρχει ένας μηχανισμός λογοδοσίας ε, και να γίνεται η αξιολόγηση από μια ανεξάρτητη αρχή και να προβλέπεται αποζημίωση και αποκατάσταση. Ε, θα μπορούσα να μπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν έχουμε χρόνο, αλλά συμπερασματικά θέλω να επιμείνω σε κάποια πράγματα που είπα πριν για το σεβασμό, την προστασία και τον έλεγχο και θέλω και να σας ενθαρρύνω να δείτε ότι το πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί τη βάση, όχι την οροφή, δηλαδή είναι το ελάχιστο. Δεν σημαίνει ότι ε, αρκεί να φροντίσουμε να μην βασανίζεται ένα παιδί ή να μην ξέρω πρέπει να δούμε και το θέμα της αξιοπρέπειας των ανθρώπων αυτών. Μόνο τότε συνάδουμε με τόσα λένε οι συνθήκες και τόσα λέει και το άρθρο 21 που πρέπει να το κοιτάτε κάθε τόσο και να το λαμβάνετε υπόψη σας στις διεθνείς συνεργασίες τις οποίες καταλήγετε με τρίτες χώρες ώστε να είστε σίγουροι ότι αποδέχονται όλες αυτές τις αρχές και αυτές οι τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Δύο έχουν ζητήσει το λόγο, Λαμπέρ και Μπερτζιά. Δεν ξέρω αν και κάποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Η Τζιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω... Δεν θα κάνω πολλές ερωτήσεις, λίγες. Πρώτα απ' όλα, ε, έγινε αναφορά νομίζω ε, σε αρκετές ομιλίες ε, στο θέμα του, της ταυτοποίησης όταν γίνεται η προετοιμασία για την επιστροφή. Ξέρουμε ότι τα πράγματα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα κατά πόσον όλα τα κράτη-μέλη έχουν και μία διαδικασία περί απάτριδων. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το επιχείρημα που προβάλλεται από τη στιγμή, ας πούμε για τους Ροχίνγκα. Αν είναι κανείς Ροχίνγκα από το Μπαγκλαντές, δεν είναι κανείς υπηκός του Μπαγκλαντές, ενώ πολλές φορές καταγράφεται ως τέτοιος. Κατ' ουσίαν είναι κανείς άπατρης. Γι' αυτό λοιπόν ε, ρωτώ, τα κράτη-μέλη έχουν τέτοιου είδου διαδικασίες που να λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα ουσιαστικά προβλήματα. Ίσως να μην είναι τα σημαντικότερα, αλλά είναι και αυτά πραγματικά προβλήματα. Κατόπιν, όσον αφορά ε, τις ίδιες επιστροφές. Ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ελέγχει ε, τις πτήσεις και τα αεροσκάφη. Αυτό το είχαμε θίξει όταν ασχοληθήκαμε με την οδηγία περί επιστροφών. Εσείς στο πάνελ τι πιστεύετε, τι σημαίνει επιστροφή που να είναι βιώσιμη. Υπάρχει ένα κομμάτι της διαδικασίας ασύλου όπου αν οι άνθρωποι ε, επιστραφούν, τι θα γίνει μετά υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου, να μπορεί κανείς να ελέγξει αν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση έλαβε τη σωστή απόφαση. Δηλαδή υπάρχει ένας μηχανισμός ε, συνέχειας, παρακολούθηση. Τι γίνεται, επιστρέφονται και μετά τι γίνεται. Επίσης για τις ε, προαιρετικές επιστροφές ε, και για την απαγόρευση επιστροφής έπανισόδου, αυτό είναι το τιμωρητικό στοιχείο της ε, οδηγίας ε, περί επιστροφών. Θέλω να ρωτήσω, ξέρετε μήπως ε, ποιες ήταν οι επιπτώσεις αυτής της απόφασης. Μιλήσατε για αποτελεσματικό έλεγχο. Τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Αυτά είχα να ρωτήσω και ευχαριστώ πολύ. Έχω και πολλές άλλες ερωτήσεις, αλλά ίσως να τις κάνω κάποια άλλη φορά. Ήταν, είπατε ήδη αρκετά, ρωτήσατε αρκετά Τζιν. Η Μαρή Κριστίν έχει το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους τρεις ομιλητές και ιδίως τον κύριο Λιούις. Ο τρόπος με τον οποίο άρχισε την παρέμβασή του δείχνει ότι ο ίδιος δεν είχε καμία δυσκολία να έρθει στις Βρυξέλλες, διότι κάθε φορά που μιλούμε για μεταναστευτική πολιτική, εκεί πρέπει να ξεκινούμε. Ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα, δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα στην κινητικότητα. Τα ίδια που λέγα προηγουμένω. Ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει δικαίωμα στην κινητικότητα, δύο τρίτα είναι υποχρεωμένα να μείνουν εκεί που βρίσκονται κατά απόλυτη περιφρόνηση του άρθρου 13 της Οικουμενικής Διακήρυξης Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Το άλλο που θέλω να ευχαριστήσω είναι που υπενθυμίσατε τα δικαιώματα των ανθρώπων και το σύνολο των διεθνών συνθήκων που έχουν συνυπογράψει οι χώρες μέλη μας, εκτός βέβαια από τα δικαιώματα για την επανένωση των μεταναστών με τις οικογένειές τους, που λέει ότι κάθε μετανάστης, όποιο και αν είναι το καθεστώς του, έχει τέτοια δικαιώματα. Άλλα διεθνή κείμενα υπενθυμίζουν αυτό που είναι προφανές, ότι όλοι οι μετανάστες έχουν δικαιώματα ανεξαρτήτως καθεστώτος. Έρχομαι τώρα στην πολιτική επιστροφών. Ο κύριος Λετζέρη μας είπε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα διότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στον αριθμό των προσώπων που ζητούν άσυλο και στον αριθμό των προσώπων που τελικώς τους χορηγείται το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Τι θα πει μεγάλη απόσταση. Νούμερα. Θα υπενθυμίσω νούμερα. 61% των προσώπων που ζητούν άσυλο λαμβάνουν στον πρώτο βαθμό δικαίωμα στη διεθνή προστασία. 61%. Δηλαδή σχεδόν τα δύο τρίτα. Και κυρίως αν προσθέσουμε και τα υπόλοιπα 17% που λαμβάνουν το δικαίωμα αυτό, σε παραπάνω βαθμούς δικαιοδοσία. Ε, δεν είναι πολύ, πολύ μεγάλη απόσταση. Υπάρχει όμως μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις χώρες μέλη. Από 8% κατά μέσον όρο, 8% στην Ουγγαρία. Τι περίεργο. Σε 83%, πάνω από 80% σε πολλές άλλε χώρες μέλη. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εν προκειμένου και γνωρίζω ότι δουλεύουμε όχι εγώ άμεσα, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια εναρμόνισης, αλλά δεν πρόκειται να διευθετηθούν αυτές οι πολύ μεγάλες διαφορές. Όσο δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αυτά, θα συνεχίσουν οι χώρες μας να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες του, διότι υπάρχουν ανισότητες. Και όλοι όσοι δεν λαμβάνουν το ασύλο δεν σημαίνει ότι είναι κακοί μετανάστες. Υπάρχουν ανισότητες και σε ό,τι αφορά τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης και θα συνεχίσει να παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν απευθυνόμενοι σε εσά τους δυο. Frontex και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς θα εξασφαλιστούν οι πολιτικές επιστροφών με ταυτόχρονο σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή δεν θα γίνονται συλλογικές επαναπροωθήσεις. Άκουσα τις προτάσεις που είπατε θα κάνετε στις χώρες μέλη και κάπως με ανησυχούν πώς θα εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει ατομική εξέταση της κάθε περιπτώσεως, πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων τους, πλήρης σεβασμός των διαδικασιών. δεν θα πλήξουν οι επιστροφές ευάλωτα άτομα. Πώς θα αποφύγουμε να τους επιστρέψουμε σε χώρες όπου ενδεχομένως θα υποστούν παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή του. μπορεί να υποστούν βασανιστήρια. Πάλι κατά παραβίαση των διεθνών κειμένων. Και επίση, συμφωνώ όταν λέτε ότι η διαχείριση της μετανάστευσης δεν μπορεί να περιορίζεται μονάχα σε ζητήματα πολιτικής επιστροφών. Τι θα πει όμως αυτό συγκεκριμένα για εσάς και ειδικώ για τον οργανισμό Frontex. Τι θα πει αυτό. Και τέλος, ισορροπημένη διαχείριση των επιστροφών απέναντι στην Αφρικανική Ήπειρο. Ναι, αλλά πέστε μου τι ακριβώς κάνετε εν προκειμένου. Και τέλο, και συμφωνώ με αυτά που ρώτησε προηγουμένως η Σοφή Ιντφέλτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Πώ μπορεί να διασφαλίσει ότι για την πολιτική αυτή, εμεί εδώ Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι για την πολιτική αυτή θα υπάρχει πραγματικό σεβασμό των διαδικασιών και του συνόλου των κανόνων που διέπουν τι περιπτώσει αυτέ, Η δική μα υπόθεση, η δική μα ευθύνη είναι να εξασφαλίσουμε τον σεβασμό στις διεθνεί συνθήκες. Τα λέμε αυτά σε όλα μα τα ψηφίσματα. Συγκεκριμένα όμω, τι κάνουμε για να ανταποκριθούμε στις ευθύνε μας και απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωση. Okay. Um, πολύ ωραία. Ε, 12 και 4 πρέπει να τελειώσουμε. Ε, Ω εκ τούτου, αν θέλετε να είστε λιγάκι σύντομο στι απαντήσει σα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Θα είμαι σύντομος. Η πρώτη ερώτηση αφορά τους απάτριδες και τη διαδικασία της ταυτοποίησης. Ε, οι απάτριδες επ' αυτού δεν υπάρχει πλαίσιο ρυθμιστικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από το τι ισχύει στα κράτη-μέλη που έχουν ε, τα κράτα-μέλη ε, κάποια σχετική νομοθεσία. Εμείς ε, στη διαδικασία της ταυτοποίησης δεν μπορούμε να προβούμε σε επιστροφή αν δεν γίνει αποδεκτή επιστροφή από την τρίτη χώρα αυτό είναι μια επιπρόσθετη εγγύηση. Ε, βιώσιμες επιστροφές. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να έχουμε κατά νου δύο διαφορετικά πράγματα. Πρώτον, το ότι η διαδικασία επιστροφών είναι μια διαδικασία που ελέγχεται τόσο ε, σε εθνικό επίπεδο όσο και ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί η Frontex έχει αναλάβει και αυτή κάποια συγκεκριμένη δέσμευση. Μόλις λοιπόν επιστρέψει ο, ο μετανάστης ε, στην χώρα προέλευσης, ε, γίνεται κάποια έρευνα το τι συμβαίνει μετά και τώρα αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χορηγούνται κάποια κονδύλια για τις επιστροφές. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε όσο καλύτερα μπορούμε να επενδύουμε σε κοινότητες ε, που δέχονται άτομα να επιστρέψουν. Επίσης επενδύουμε σε προγράμματα ε, τα οποία ελέγχονται για άλλους έξι ή οκτώ μήνες οι επιστρέφοντες ε, δέχονται επισκέψεις για να παρακολουθούμε και εμείς τι γίνεται τελικά. Κατόπιν, Σας είπα, στις 6 Δεκεμβρίου θα έχουμε μία συζήτηση και κλεισμένων των θυρών για τις περίφημες ε, Cheval αποστολές, Cheval Missions, ε, να δούμε πώς εφαρμόζονται οι συμφωνίες ε, στα κράτη-μέλη. Και αυτό που έχει σημασία είναι και να ξέρετε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα επηρεάσει την ερμηνεία των αποφάσεων. Τελευταία ερώτηση, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους επιστρέφοντες. Ε, είναι σημαντικό εδώ να πούμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε μαζικές επιστροφές, διότι κάθε επιστροφή βασίζεται σε μία συγκεκριμένη απόφαση, που και αυτή πάλι βασίζεται σε μία συγκεκριμένη αξιολόγηση μίας κάθε μεμονωμένης περίπτωσης. Άρα δηλαδή δεν υπάρχουν μαζικές ε, ε, επιστροφές ε, όπως το αναφέρουν κάποιοι. Και αυτές ε, οι μεμονωμένες αξιολογήσεις ε, προκύπτουν ε, και με πολύ αυστηρούς ελέγχους. Όλες οι αποφάσεις για επιστροφές περιλαμβάνουν την εμπλοκή του δικαστικού συστήματος ε, με όλες τις εγγύησεις που προσφέρει ένα δικαστικό σύστημα. Επίσης ε, υπάρχει ένα καλό δικαστικό σύστημα το οποίο θα ενισχυθεί και περαιτέρω με την ε, εντολή που έλαβε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εκτοφυλακής και Συνοριοφυλακής. Δηλαδή μας ενδιαφέρει να υπάρχει σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καλύπτεται και αυτό στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής. Εστιάζουμε ε, κατά διάρκεια των αποστολών μας ε, ε, και στο να επισημαίνουμε και διαδικασίες επί παραμπάση, κυρίως εναντίον εκείνων των κρατών που δεν εφαρμόζουν σωστά την κειμένη νομοθεσία. Κύριος Λετζέρη, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την απόσταση μεταξύ απορριφθησών αιτήσεων ασύλου και των προσώπων που ε, πρόκειται να επιστραφούν ακόμα και αν πάρει κανείς τον μέσον όρο των 61% αποδοχής εάν πάρει σε τους απόλυτους αριθμούς το 2015 σε ένα σύνολο ενός εκατομμυρίου προσώπων βλέπει κανείς ότι η διαφορά φτάνει τα 400.000 άτομα άρα είναι μια ανισχυτική κατάσταση όταν άνθρωποι δεν έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα σε παραμονή, άρα ούτε δικαίωμα σε εργασία και επομένως τελικά μια κατάσταση η οποία δεν πλαισιώνεται ορθά στις χώρες μέλη όπου βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Σε ό,τι αφορά, όπως είπε και ο Ρωσός της Κομισιόν, την συνέχεια που δίνεται στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, υπενθυμίζω ότι υπάρχει κώδικας διοντολογίας του οργανισμού μας, συνοριοφυλακής ακτοφυλακής για τις επιστροφές και ότι η αναγνώριση της κατάστασης των προσώπων αυτών από άψη κλπ. Ε, συμπεριλαμβάνεται. Το 2017 ο οργανισμός ανέπτυξε 86 αξιωματούχους παρακολούθησης και η πολιτική του οργανισμού είναι ότι όταν οι χώρες μέλη δεν είναι σε θέση να διαθέσουν εθνικούς αξιωματούχους για να ασκούν την παρακολούθηση αυτή, λαμβάνει από την δεξαμενή των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Και η διάκριση που γίνεται ανάμεσα πτήσεις που θεωρούνται πιο ευαίσθητες, δηλαδή με προορισμό χώρες οι οποίες απέχουν από τα δικά μας πρότυπα και ιδίως σε ό,τι αφορά τον σεβασμό μιας σειράς αρχών φροντίζουμε στα αεροπλάνα αυτά να βρίσκονται ε, αξιωματούχοι που παρακολουθούν την εξέλιξη των διαδικασιών. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τον οργανισμό συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Οι χώρες με τις οποίες έχουμε διεθνή πολιτική συνεργασία πιο είναι οι χώρες βέβαια με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει ιδίω σύμφωνα, compact, μέσα στα πλαίσια των οποίων γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, ε, έστω και αν είναι εκτός πλαισίου εντολής του οργανισμού μας, υπάρχουν άλλα, ε, άλλοι μηχανισμοί που επιτρέπουν την αναπτυξιακή συνεργασία. Ευχαριστώ εσείς κύριε Λιούις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομη απάντηση σχετικά με το ζήτημα της βιωσιμότητας. για την αρχή της ε, απαγόρευσης των βασανιστήριων κλπ. Εμείς ε, συζητούμε στο γραφείο μας τι ακριβώς σημαίνει η βιωσιμότητα από την άποψη των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θα εκδώσουμε κατευθυντήρες γραμμές. Είπαμε κάτι σχετικά σε αρχές και κατευθυντήρες γραμμές για τη μετανάστευση και τους μετανάστες σε ευάλωτη κατάσταση. Λέμε στις γραμμές αυτές ότι βιωσιμότητα σημαίνει ότι όταν ένα πρόσωπο επιστρέφεται θα πρέπει να απολαμβάνει ένα ελάχιστο ανθρώπινων δικαιωμάτων, δηλαδή κοινωνική προστασία, το δικαίωμα σε αξιοπρεπή εργασία, δικαίωμα σε αξιοπρεπή διαβίωση, πρόσβαση σε δικαιοσύνη κλπ. Σε χώρες όπου αυτό αυτά τα θεμελιώδη δεν είναι εξασφαλισμένα, δεν μπορεί να υπάρχουν επιστροφέ. Κάποιε άλλε πρακτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβητούν ορισμένα από τα βασικά αυτά θέματα. Και μιλώ και για κυβερνήσεις με τις οποίες διαπραγματεύεστε ανεπίσημες ε, συμφωνίες, όπως με τη Λιβύη για παράδειγμα. Πώς μπορεί να θεωρηθεί, να θεωρηθεί η Λιβύη επαρκής εταίρος ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ε, επιστρεφομένων. Και θα υπάρχουν και άλλες χώρες. Και αυτό τώρα για αυτές τις mass deportation, τις μαζικές μετακινήσεις, εννοούσα δηλαδή μεγάλο αριθμό, όχι βεβαίως συλλογικές επαναπροωθήσεις, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Μιλώντας για μαζικές εννοούσα ότι είναι μεγάλη η αριθμή ανθρώπων που θα πρέπει να επιστρέψουν και δεν έχουν δικαίωμα παραμονής. Αυτό εννοώ. Όταν μιλεί κανεί για επιστροφή τόσων πολλών ανθρώπων, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά ίσως διότι εξετάζεται το δικαίωμα του ασύλου σαν μόνο ε, δικαίωμα που επιτρέπει την παραμονή. Ενώ πρέπει να υπάρχουν και άλλα δικαιώματα που να είναι εξασφαλισμένα. Και οι επιστροφέ δεν μπορεί να είναι μόνη επιλογή. Θα πρέπει να υπάρχουν και άλλες λύσεις που να είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και πολιτικά και στην πράξη. Χωρί να οδηγούν σε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Χωρίς να σημαίνει πάλι αυτό ότι δεν μπορείτε να επιστρέφετε κανένα. Αλλά μιλώντας όπως είπα πριν για μεγάλους αριθμούς επιστροφών με κάποιο στοιχείο εξαναγκασμού ε, στις επιστροφές αυτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τους τρεις σας. Και ευχαριστώ και τους συναντέλφους για τις ε, πολύ καλές ε, παρεμβάσεις τους. Και θα τα πούμε στις 2.30. Ευχαριστούμε πολύ.